Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι έχετε επιστρέψει από το Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, Σα καλωσορίζω θερμότατα στη σημερινή μα συνεδρία. Έχετε παρατηρήσει για τη μέση διάταξη? Όχι. Στην ανακοινώσει του Προέδρου έχω μια παρατήρηση να κάνω. Boris Nemtsov war auch... Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ο Μπόρις Νεμτσόφ είχε έρθει και εδώ στην Επιτροπή μα Την τελευταία 15 ετία προσωπικά είχα αμέτρητες συζητήσει μαζί του στη Μόσχα, στο Στρασβούργο, στη Βρυξέλλε και αλλού. Και έμαθα να τον εκτιμώ ως ειλικρινή άνθρωπο, πάρα πολύ χαρισματικό και με τεράστιο θάρρος. Είχαμε συζητήσει και για τη προσωπική του κατάσταση, του κινδύνους που διέτρεχε και είχε πλήρη επίγνωση αυτών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η δημοκρατική πλέον αντιπολίτευση στη Ρωσία έχει χάσει ένα φάρο της και αυξάνεται όλο και περισσότερο κίνδυνος να πέσει ένα πέπλο πάνω από τη Ρωσία δεν ξέρω ποιος ευθύνεται προσωπικά, αλλά όλο και περισσότερο το σύστημα που εξελίσσεται σε αυταρχικό και αυτοκρατορικό φέρει ευθύνη. Ακούω από τις διοκτικές αρχές διάφορες σκοτεινές θεωρίες συνωμοσία και οι νεκροί και οι κρατούμενοι αυτοί που είναι στα γκουλάκ του Πούτιν ή που έμειναν εκεί. Πάντα όλους τυχαίως ήταν αντιφρονούντες, αντικαθιστοτικοί και άνθρωποι επικίνδυνοι για το σύστημα και ουδείς άλλος. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν φαίνεται ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Μπορίς Νέμτσοφ είχε δηλώσει ότι είχε αποδείξεις για την άμεση ανάμειξη της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και μάλλον και αυτό δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για ορισμένου κύκλους που φέρουν και ευθύνη. Θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μπορίς Νέμτσοφ, και ταυτόχρονα θα σας παρακαλούσα παντού και στη Ρωσία να υποστηρίζουμε τους δημοκράτες και όσους είναι υπέρ των δημοκρατικών αξιών και αρχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 4 μια συζήτηση με τον κύριο Κρέχενμπουλ. Μάλλον Βόρεια Γερμανία θυμίζει αυτό το όνομα σας παρά Ελβετία. Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας Αρρωγή και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή, επικεφαλής της UNRWA. Επανειλημμένα είχαμε και εκεί συζητήσεις και σε σχέση με τις εξέλιξεις στο Παλαιστινιακό Παλαιστίνη-Ισραήλ και πάλι είναι βαθιά η ανησυχία μας για τις εξελίξεις εκεί λόγω της έλλειψης οτιδήποτε οικονομικής προοπτικής. Και αν δούμε τι γίνεται στη Γάζα και το ρόλο που παίζει η Χαμάς και σε σχέση με τα όσα γίνονται στη Δυτική Όχθη θα σας παρακαλούσαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε την κατάσταση, ε, να μας παρουσιάσετε πώς έχει και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε εμείς να δραστηριοποιηθούμε για να βοηθήσουμε. Γιατί οπωσδήποτε και εκεί πάντα χρειάζεται έλεγχος, γιατί ρέουν πάρα πολλά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καμιά φορά ε, μας λυπεί το γεγονός ότι δεν προβάλλεται αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται αρκετά ορατό αυτό. Ε, Ενδεχομένω να αφαιρθείτε και σε αυτό. Πάντως θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα, να πιάνει τόπο αυτή η βοήθεια και να ενισχύσει και την πολιτική διαδικασία. Κάτι να γίνει, να υπάρξει η δυνατόν πολιτική ε, ειρηνική επίλυση. Οι πρόσφυγες είναι και στην γειτονία ε, των χωρών αυτών και είναι και επικίνδυνα τα πράγματα. Τις περασμένες μέρες πήγαμε μια αντιπροσωπεία στο Λίβανο και στην Ιορδανία προσωπικά και στο Ιράκ πήγα, στο Ερμπίλ και στη Βαγδάτη και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να ειδωθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ε, πάντα, επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει και για το Λίβανο και για την Ιορδανία. Είναι πάρα πολλοί οι Σύριοι πρόσφυγες που τώρα καλούνται να ε, περιθάλψουν και να φροντίσουν και βοηθάει και η ΟΡΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε ε, και να δούμε ότι υπάρχουν και Παλαιστίνοι πρόσφυγες εκεί. Στο Λίβανο ε, μας λένε ε, ότι δεν θα φτιάξουμε καταβλισμούς για τους Σύρους γιατί ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Γιατί έχουμε ακόμα 200-300 χιλιάδες Παλαιστινίους πρόσφυγες σε καταβλισμούς εδώ και 60 χρόνια. Οπότε για τους Σύρους δεν φτιάχνουμε. Έχετε το λόγο να μας τα παρουσιάσετε όλα αυτά και να μας τα εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Πολύ σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και ιδίω για την ευκαιρία να αντιμετωπίσω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για την στεναρή και ανατρέχουσα στο βαθύ παρελθόν υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ούνερα, προς την ε, υποστήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων στη Μέση Ανατολή. Να σας ευχαριστήσω για την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τα μεμονωμένα κράτη-μέλη που μας έχουν δώσει την απαραίτητη υποστήριξη στο φορέα μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας έχει δώσει για να μπορέσει να υπάρξει η σωστή υποστήριξη. Αυτό περιλαμβάνει την οικονομική αρρωγή για του Παλαιστινίου πρόσφυγες και για την Ούνορα και επίσης και για το ψήφισμα του 2014 για τη Γάζα, τη σημαντική ψηφοφορία για το ε, κρατικό καθεστώς της Παλαιστίνης και επίσης για το ψήσιμο για την οικονομική κατάσταση Σούρα που το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα και θέλω λοιπόν να εκφράσω την αναγνώρισή μου για τη συζήτηση που διεξαγάγατε για το θέμα αυτό και τη σημασία που επέχει για μας. Θα ήθελα να αντιμετωπίσω μερικές πτυχές της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ιδίω τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει αντίκτυπο για τις κοινότητε των Παλαιστινίων προσφύγων. Πρέπει να σας πω ότι έρχομαι ενώπιόν σα σε μια εποχή με μεγάλες ανησυχίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιβεβαιώσω αυτό. Ξέρετε ότι η περιοχή είναι σε μια εποχή ταραχώδη και δύσκολη, μια εποχή η οποία σημαδεύεται από τη συνέχιση της κατοχής και του αποκλεισμού της Γάζας, της στρατιωτικής αντιπαράθεσης που είδαμε και το καλοκαίρι στην περίπτωση της Γάζας, αλλά και την βαθιά αντιπαράθεση που συνεχίζεται στη Συρία και που έχει σημαντικό αντίκτυπο και στις όμορες χώρες. Από τη δική μας οπτική γωνία βλέπουμε στον πυρήνα όλων αυτών των προβλημάτων την απουσία μιας πολιτικής λύσης στα προβλήματα της περιοχής. Ως αποτέλεσμα αυτής της απουσίας συνεχίζεται με αδίδυτο τρόπο η ριζοσπαστικοποίηση στην περιοχή και οι διάφορες μορφές εξτρεμισμού σε όλη τη Μέση Ανατολή, κάτι που έχει σημαντικές επιδράσεις στις κοινότητες που προσπαθούμε εμείς να βοηθήσουμε. Συγχρόνως και λόγω της αντιπαράθεσης αυτής βλέπουμε να αποδυναμώνονται οι κρατικοί θεσμοί στην περιοχή. Οι κυβερνήσεις λοιπόν οι κυβερνήσει που υποδέχονται του πρόσφυγε είναι φυσικά η κύρια εταίροι τη ούρα για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων. για να παρουσιάσουμε την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Όπω ξέρετε σε όλη την Πρόσω Ανατολή υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες που υποστηρίζονται από την Ούντρα. Είναι το ίδιο με τον πληθυσμό της Νορβηγίας ή με την Σιγκαπούρη. Αλλά φυσικά δεν έχουν εστίες, δεν έχουν χώρα δική τους και εξαρτώνται απόλυτα από την υποστήριξή της Ούρα. Στην Δυτική Όχθη η κατάστασή τους είναι μια κατάσταση που προσδιορίζεται από τη συνέχιση των επικισμών του Ισραήλ, από τη βία που ασκείται από τους επικιστές, περιπτώσεις καταστροφής και ανατίναξης οικειών και από άλλα γεγονότα τα οποία οδηγούν στον κίνδυνο της ε, βίαιης μετατόπισης και εκένωσης κοινοτήτων Βεδουίνων. Είναι λοιπόν μια συνεχής αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Βλέπουμε στη Δυτική Όχθη ένα πρόσθετο φαινόμενο που έχει μεγάλες συνέπειες, είναι η παρακράτηση των φορολογικών εσόδων. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις στους φορείς και τους θεσμούς της Παλαιστινικής Αρχής. Μειώνεται η ικανότητα δράσης της. Υπάρχει μια βαθμία μετάφορα των ε, απαιτήσεων και των αναγκών του πληθυσμού προς την κατεύθυνση της ούρα που καλείται να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες. Βλέπουμε λοιπόν πολύ περιορισμένη δυνατότητα ικανοποίηση αυτών των αναγκών από την Παλαιστινική Αρχή. Στη Γάζα φυσικά ξέρετε τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι. αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση ουσιαστικά επιβίωσης για τον πληθυσμό της Γάζας. Μια υπαρξιακή κρίση. Είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα των ενεργειών που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, του αποκλεισμού της Γάζας και των επιπτώσεων που προέγγιψαν για το λαό της Γάζας. Να σας δώσω μερικούς δείκτες μονάχα. Το 2000 όταν η κατάσταση δεν ήταν φυσιολογική, αλλά τουλάχιστον ήταν πιο ανοιχτή σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία στη Γάζα. Είχαμε 80.000 Παλαιστίνιους που βασιζόταν στην επιστηστική βοήθεια της ούρα στην λοριδά της Γάζας. Σήμερα, μετά από τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί, έχουμε πάνω από 860.000 άτομα που εξαρτώνται από τα τρόφιμα της ούρα δεν προσπαθώ με τα στοιχεία αυτά να σας δείξω πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία μας να προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σας τα λέω αυτά τα στοιχεία γιατί σας το παρουσιάζω αυτό σαν μια στατιστική όνειδος, ντροπή. Όταν από 1,8 εκατομμύρια 860.000 βασίζονται στην επιστημιστική βοήθεια της ούρα και εδώ δεν αναφέρω αυτούς οι οποίοι βασίζονται στο παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων, το WFP. Ο λόγος για τον οποίο είναι έτσι η κατάσταση είναι γιατί οι επιχειρηματίες που είχαν τις δικές τους επιχειρήσεις εκεί έδιναν απασχόληση, κάνανε εξαγωγές στο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη και στην Ευρώπη ακόμα. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, έχουν καταστραφεί, αναγκαστήκανε να απολύσουν το προσωπικό τους, χάσανε ακόμα και τα σπίτια τους πολλές φορές και ζουν σε δωμάτια τα οποία είναι νοικιασμένα όπως όπως και ζουν, επιβιώνουν με τη βοήθεια της ούρα. Αλλά μιλάμε για ένα πληθυσμό ιδιαίτερα μορφωμένο. Ο πληθυσμός Γάζας είναι ιδιαίτερα μορφωμένος και με, με σημαντικά προσόντα και θέλουν μόνοι τους να υπομισθούν την προστασία και τη διατροφή της οικογένειάς τους. Δεν θέλουν να εξαρτώνται από την ούρα. Ούτε αυτοί, ούτε εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση πραγμάτων. Θέλουν να ξανανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και τα μαγαζιά τους, να ξαναρχίσουν να εξάγουν, θέλουν να είναι τμήμα της κοινότητας στην οποία ζουν, θέλουν να δουν τα βασικά προβλήματα της κατάστασής τους να αντιμετωπιστούν. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει και τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφαλειά του, που φυσικά είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για τη Γάζα. Ήδη οι συνθήκες του αποκλεισμού σημαίνουν έλλειψη ελευθερίας κίνησης, διακίνησης, ελάχιστες δυνατότητες απασχόλησης, αλλά επιπλέον έχουμε και την πολεμική σύγκρουση του περασμένου καλοκαιριού με την τεράστια καταστροφικότητα που είχε, η οποία ήταν χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Γάζας τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε μοναχά τα άτομα τα οποία είναι άνεργα, αλλά έχουμε 100 με 125 άστεγους στη λόριδα της Γάζας μετά από την καταστροφή που έγινε στον πόλεμο, την απώλεια των αισιών τους και οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει λένε ότι 96.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί τελείως ή έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες άλλων κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρέ ζημίε. 20.000 αυτέ που έχουν υποστεί σχεδόν ολοκληρωτικέ. Έχουμε λοιπόν τις, ε, τα προβλήματα αυτά, του άστεγου και έχουμε και το συνολικό τραύμα που νιώθουν οι άνθρωποι τη Γάζα. Παρόλο που 540 παιδιά σκοτώθηκαν στην, ε, στις πολεμικές επιχειρήσεις πέρσι, πολλά από αυτά κάτω από την ηλικία των 12, 40%, 70% συγγνώμη. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν γύρισαν στα σχολεία τους. Πάνω από χίλια παιδιά θα, που έχουν τραυματιστεί θα έχουν μόνιμες αναπηρίες στη λόγια της Γάζας. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο το τραύμα από την καταστροφή των οικειών και των κτηρίων. Είναι και ο αντίκτυπος σε ανθρώπινους όρους στην κοινότητα της Γάζας. Και ενώ σήμερα εστιάζουμε στην ε, βραδία διαδικασία ανοικοδόμησης στη Λόριδα της Γάζας και προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό εξουσίας επίσης στη Γάζα και το γεγονός ότι η κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να μπορέσει να αναλάβει απόλυτα τα ενία της εξουσίας στη Γάζα. Αντιμετωπίζουμε επίσης και το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης και του γεγονότος ότι πολλές από τις υποσχέσεις που δόθηκαν στη συνδιάσκεψη του Κάιρου δεν έτυχαν συνέχεια. <clears throat> Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο όμως είναι ότι εν, ενδιαμέσως έχετε μια κοινότητα στη Γάζα και μια κοινότητα στο Ισραήλ που ζουν πλάτη με πλάτη η μία με την άλλη. Είναι γενιές νέων που μεγαλώνουν χωρίς την παραμικρή επαφή, χωρίς να ξέρουν τι ζει η άλλη πλευρά. Μου το έλεγε ένας επιχειρηματίας 58 χρονών στη Γάζα πέρσι, μου έλεγε ότι τα παιδιά του δεν ήταν τόσο κοντά στο Ισραήλ όπως ήταν ο ίδιος. αυτό είχε μεγαλώσει σε επαφή με Ισραηλινούς, είχε αντιμετωπίσει Ισραηλινούς στην επιχειρηματική του ζωή, είχε εμπορευτεί μαζί τους, είπε πολλές φορές διαφωνώ μαζί τους αλλά νομίζω ότι ακόμα μπορώ να καταλάβω τη λογική τους και τον τρόπο με τον οποίο βρέμουν τα πράγματα. Τα παιδιά μας όμως είπε, δεν έχουν ποτέ συναντήσει ένα Ισραηλινό στη ζωή τους. Δεν τους έχουν δει ούτε από μακριά. Υπάρχει μια πραγματικότητα απόλυτου διαχωρισμού. Ζουν πίσω από τύχη, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Πρόσφατα ένα έγγραφο στο New York Times έλεγε 42% των Ισραηλινών δεν είχαν ποτέ συναντήσει ένα Παλαιστίνιο. Μα αυτό δεν μπορεί να είναι μια βάση για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στο μέλλον. Και θα επανέλθω στο θέμα της Συρίας και των περιφερειακών συνεπειών που προκύπτονται. Ένα μεγάλο μέρος της εστίασης της Ευρώπης και ημών με ύψιλον ε είναι στην ασφάλεια της Μέση Ανατολής. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια σαφή σύνδεση σε περιφερειακό επίπεδο και ότι οι νέοι της Γάζας, 65% του πληθυσμού της Γάζας είναι μικρότεροι από 25 ετών, αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα. Είναι άνθρωποι που είναι μορφωμένοι, που δεν είχαν καμία ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον να το πράξουν. Το θέμα της Συρίας φυσικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχουμε καταγράψει με μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση για την Συρία και το Ιράκ που παρουσιάστηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Είναι ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα, μία από τις πιο καταστροφικές σειράξεις που έχουμε αντιμετωπίσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 95% του πληθυσμού των Παλαιστινίων προσφύγων που ήταν στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης γιατί ήταν τμήμα της οικονομίας και της κοινωνίας της Συρίας, σήμερα εξαρτώνται απόλυτα από την ώρα. 60% των προσφύγων στη Συρία από την Παλαιστίνη ήταν 550.000 πριν από τον πόλεμο, τώρα έχουν μετακινηθεί, έχουν εκτοπιστεί είτε εσωτερικά ή έχουν αναγκαστεί να φύγουν σε άλλες χώρες. 44.000 στο, στο Λίβανο, 14.000 στην Ιορδανία, 4.000 στην Αίγυπτο και 4.000 στην Τουρκία, μεταξύ άλλων πολλές από τις εγκαταστάσεις μας έχουν καταστραφεί ή υπό σημαντικές ζημίες. 6 από 219 σε όλη τη χώρα, οι οποίες τρέχουν έχουν ε, δηλαδή η καταστροφή κατά τη διάρκεια της μικρουσίας και όλα αυτά χωρίς να παραλείψουμε το ποιες είναι συνέπειες για τις όμορες χώρες, Λίβανο και Ιορδανία, εκεί όπου ήδη έχει μετακυριστεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του βάρους των ε, ε, των προσφύγων ε, των Παλαιστινίων ιστορικά και τώρα και από τη Συρία. Οπότε πρέπει να σας τονίσουμε το ότι αυτές όλες οι Παλαιστίνες κοινότητε στην Μέση Ανατολή, όλες οι κοινότητες αυτές αντιμετωπίζουν μια κρίση προστασίας. Και επίσης αυτό έχει να κάνει και με το πόσο ευάλωτη είναι και οπότε συνεχώ νιώθουν όλα περισσότερη απογοήτευση για την καταστασή του θεωρούν τους έχουμε εγκαταλείψει, του έχουμε ε, ξεχάσει ε, στα πλαίσια του, του, του διεθνούς σκηνικού όπως διαμορφώνεται η Ούνρα, η Ούνρα. Τώρα τι κάνει. Θα ε, συνδυάσουμε τον Μάιο, γιατί είπαμε ότι πρώτη 65 χρόνια λειτουργία μα που κλείνουμε. Οπότε θα πρέπει και να σας τονίσω σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα 65 χρόνια λειτουργία τη Ούνρα σημαίνει κατά τη γνώμη μου δύο τεινά εκτός άλλων σημαίνει ότι έχουμε βρει διάφορους τρόπους να μπορέσουμε να παράσχουμε ε, χρήσιμη ε, βοήθεια, να μπορέσουμε να παράσχουμε πολύτιμες ε, υπηρεσίες σε αυτές τις μεγάλες κοινότητες των προσφύγων. Όμως, σημαίνει όμως ότι όταν τα κάποια θέματα δεν αντιμετωπίζονται από την πολιτική πτυχή τους και δεν υιοθετούνται πολιτικές λύσεις, τότε τότε προκύπτουν αυτά τα 65 χρόνια λειτουργία τη Τσούνα, γιατί ποτέ δεν είχε κανεί προβλέψει ότι θα παραμείνουμε εν λειτουργία επί τόσο χρόνο. Οπότε απουσία πολιτική λύση, τελικά αυτό ε, σήμαινε ότι εμεί θα παραμείνουμε σε λειτουργία για τόσα χρόνια και, και άλλα. Πριν από 11 μήνε μόλι μπήκα στην υπηρεσία, οπότε να σα πω τι διαπίστωσα. Τι με εντυπωσίασε. μια που είχα πριν δουλέψει 20 χρόνια στα πλαίσια του Ερυθρού Σταυρού. Είναι αξιοπερίγοντο τι σημαίνει στην ώρα γιατί συνδυάζει ανθρωπιστικό ρακτήρα ε, αποστολές και από την άλλη μεριά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και θα πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο πέτυχε η Ινουρα για την ανάπτυξη είναι ε, ένα ρεκόρ παγκόσμιο ούτως είπε να ρίξετε μια ματιά τι έχει γίνει παντού. Γιατί κοιτάξτε προσεκτικά από πλευρά υγεία, από πλευρά εκπαίδευση. Ε, τι, τι επιδόσεις έχουμε πετύχει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε συμβάλει όσον αφορά την ανάπτυξη του, των ανθρωπίνων πόρων, του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Και αυτό μου το λένε παντού όπου πηγαίνω. Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε εδώ τι δύο όψει του νομίσματο όσον αφορά το Παλαιστινιακό. Από τη μια μεριά έχουμε αυτή την ιστορία απογοήτευση, ε, απώλεια, εγκατάλειψη, όλα αυτά τα οποία του κάνουν να αισθάνονται θύματα. Από την άλλη όμω έχουμε και όλα αυτά που έχουν πετύχει οι Παλαιστίνοι με τι προσπαθίε στα πλαίσια τη παιδεία και σε συνεργασία με την Ούνουρα, αλλά όχι μόνο. Αυτό ήθελα να σα αναφέρω οπωσδήποτε. Επίσης, είναι σαφές ότι έχουμε πολλαπλές προκλήσεις. Δηλαδή ότι αυτά τα οποία έχουμε πετύχει στον τομέα της παιδείας και της υγείας είναι επιδόσεις αντιστρεπτές. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις συγκρούσεις γύρω-γύρω. Έχουμε τη Συρία. Έχουμε ε, αυτό το, τον αποκλεισμό στην Γάζα. Οπότε βλέπετε ότι κάποια στιγμή όλα όσα έχουμε πετύχει σε υγεία και παιδεία είναι δυνατόν να αντιστραφούν, να γκρεμιστούν. Οπότε και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την Συρία, να βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους πρόσφυγες από την ε, Συρία σε Λίβανο και η Ιορδανία. Όμως μη θεωρείτε το ότι δεν υπάρχουν απώλειες. Έχουμε χάσει 14 ε, συναδέλφους στην Συρία, 25 αγνοούμενοι, και άλλοι 11 πέρσι στην Γάζα. Να τι γίνεται όταν κανείς δουλεύει στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Τώρα έχουμε και άλλη μια πρόκληση να αντιμετωπίσουμε ότι δηλαδή οι αιτήσεις δαπάνες μας για παιδεία, υγεία και τις άλλες ανάγκες είναι 1,2 δις αμερικανικά δολάρια. Φυσικά είναι σοβαρό ποσό που πρέπει κανείς να κινητοποιήσει και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί δανειστές, δωρητές ας πούμε στο έργο της Ούνρα. Οπότε έτσι προβάλλεται το έργο μας και είναι σημαντικό να διαπιστώνετε το τι πετυχαίνουμε. Βέβαια υπάρχουν και κάποια κενά και ένα από αυτά είναι πολύ οδυνηρό. Με εξέπληξε όταν διεπίστωσα ότι γίνεται τέσσερις μήνες μετά τη διάσκεψη του Καΐρου θα έπρεπε να διακόψουμε ελήψη χρημάτων τα όσα κάναμε για τις επισκευές των καταβλισμών στην Γάζα. Από Γερμανία και Σαουδική Αραβία υπήρχαν κάποια χρήματα αλλά ξαφνικά τελειώσανε. Οπότε τώρα θα πρέπει να τρέξουμε, να πασχίσουμε, να βρούμε για αυτές τις επισκευές των καταβλισμών περισσότερα χρήματα. Και εσείς δείτε για σταθερότητα και ασφάλεια αλλά και μετανάστευση. Οπότε πρέπει να σας πω ότι οι πρόσφυγες οι Παλαιστίνοι από την Συρία που προσπαθούν να πάνε κάπου αλλού και κυρίως στην Ευρώπη είναι όλο ένα και περισσότεροι. Γι' αυτό και ε, είναι περήφανοι από τη Γάζα που μπορούν να φύγουν για να πάνε να βρουν εναλλακτικέ. Πάντω αυτό από πλευρά οικονομική θα έχει άμεση συνέπειε για όλου. Εκεί. Τώρα, κλείνοντα, Πρόεδρε, θα πρέπει να σας πω κάτι δηλαδή, για αυτή την συνεχή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας τονίσω ακριβώς ποια είναι η σημασία της. Διπλωματική και πολιτική δέσμευση, αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Εγώ εκπροσωπώ αυτόν τον φορέα που δίνει τη μάχη του στο ανθρωπιστικό τομέα και στην ανάπτυξη και είναι ό,τι πιο σημαντικό σήμερα και για τους Παλαιστίνιους και για όλη την περιφέρεια. Γιατί όταν υπάρχει κάποιο είδου πολιτική δέσμευση τόσο ώστε κανείς να χτυπήσει τις ρίζες του φαινομένου, της αιτίας αυτών όλων των εξελίξεων που αφορούν την περιοχή. Άρα θα πρέπει να γίνεται διάλογος, διάλογος μαζί σας, διάλογος με τα μπλεκόμενα μέρη εκεί, με όλους τους μπλεκομένους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχιστεί αυτό το πολιτικό γίγνεσθε και επίσης έτσι να επισκέπτεστε στην περιοχή. Όπως το έχετε ήδη κάνει, εμείς ε, ευχαρίστως πάντοτε ε, στηρίζουμε τις προσπάθειές σας για να μπορείτε και εσείς να δείτε επιτόπου τι γίνεται, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ήμασταν ε, ουσιασμένοι με το ότι η κυρία Μογκερίνη έκανε το πρώτο της ταξίδι εκτός εκεί. Πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο έστειλε. Πήγα μαζί της στη Γάζα. Χρειάζεται τέτοιου μηνύματα να παίρνει η περιοχή εκεί. Επίση, έκκληση έχω και προ εσά να συνεχίζετε να μα υποστηρίζετε ω ε, φορέα. Πολλέ φορέ λένε ε, κάποιοι 65 χρόνια πέρασαν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, φυσικά μα να μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν είναι το θέμα η ονορά. Το θέμα είναι η περιοχή αυτή, η ειρήνη, η σταθερότητα, η ειρηνική συνύπαρξη του κόσμου. Οπότε και εμεί τώρα Είμαστε ένας από τους αξιόπιστους παράγοντες και εμπλεκομένου. Μπορούμε να παράσχουμε πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε αυτήν την τόσο ευάλωτη κοινότητα. Όμως, στόχος μας δεν είναι να είμαστε εκεί αενάως. Αν μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Άρα χρειάζεται πολιτική δέσμευση, χρειάζεται ε, θεσμική υποστήριξη προς ούνρα για το έργο μας και από πολιτικής και οικονομικής απόψεως. Πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος, δυστυχώς. Gracias. Κυρία Βαλενσιάνο, ευχαριστώ. Δύο πράγματα ήθελα να πω. Πρώτον, Πρόεδρε, σε σχέση με τα όσα εισαγωγικά είπατε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία στη Ρωσία. Θα πρέπει να διατρανώσουμε, πιστεύω, εδώ στην Επιτροπή μας ότι απαιτούμε άμεση όσο και αποτελεσματική διερεύνηση. Γιατί ήδη είναι πολύ η ε, Ρώσοι ε, αντιφρονούντες και αντικαθιστοτικοί που έχουν δολοφονηθεί χωρίς να εξηχνιαστεί η δολοφονία. Θα πρέπει να καταλάβει η Ρωσία ότι περιμένουμε οπωσδήποτε να χυθεί άπλετο φως. Και σε σχέση με την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε, θα ήθελα να σας υποβάλω την εξής ε, σκέψη. Γιατί εξηγήσατε ποια είναι η οικονομική ασφυξία, η ηθική και πολιτική ασφυξία, στην οποία έχουν υποβληθεί οι ε, Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Και τα είδαμε όσοι πήγαμε εκεί στην περιοχή διεισόμαση. Αλλά δεν πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο εμείς όλοι μαζί τροφοδοτούμε το σύστημα. Από τότε που η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρηματοδοτεί ανοικοδόμηση στη Γάζα ε, και νοσοκομεία και την ίδια και την ούρα και η ούρα πολύ λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε αλλά αυξάνει πάντα τη χρηματοδότηση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά τι κάνει συνεισφέρει στη διατήρηση του status quo. Διότι όσα λεφτά και να στείλουμε, η Ισραηλινή πολιτική συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι εμείς χρηματοδοτούμε. Και εμείς το ξαναχρηματοδοτούμε από την αρχή μετά. Έτσι είναι φαύλος κύκλος 50 ετών. Είναι προφανές ότι θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε και να βοηθούμε τους Παλαιστινίους οι οποίοι βρίσκονται στη δινή κατάσταση στην οποία περιγράφεται. Αλλά το επόμενο βήμα τώρα ποιο θα πρέπει να είναι έτσι ώστε ουσιαστικά να μην γινόμαστε συνένοχοι ενός status quo που καθημερινά επιδεινώνεται όσο διαρκεί, πάνω από 60 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά της ώρα, την οποία τιμώ και σέβομαι τα μάλα. Ja, dankjewel. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φώτσμαν, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για το φόρο τιμής που αποτίσατε στο συνάδελφο πολιτικό Μπορίς Νέμτσοφ, ο οποίος δολοφονήθηκε. Ο Μπορίς πέθανε για τη δημοκρατική του δράση. Και όπως και προλαλήσασα, θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να ζητήσω ε, και η ε, Επιτροπή μας να απαιτήσει ανεξάρτητη διερεύνηση αυτής της δολοφονίας. Εμείς στο Κοινοβούλιο και εδώ στην Επιτροπή μας είμαστε κατεξοχήν αρμόδιοι για να εκφράσουμε αυτή την έκκληση. Επανέρχομαι και ε, στην ώρα που είπατε ότι 65 χρόνια δράση έχετε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και να σας συγχαρώ. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας, ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες συχνά και έχετε αποδείξει ότι ο φορέας σας επίσης έχει χάσει και ε, εργαζομένους επί έχουν αφήσει τη ζωή τους εκεί και θα πρέπει και εμείς να εκφράσουμε την αναγνώρισή μας και να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επί κάνουν τέτοια σκληρή δουλειά σε τέτοιες ε, συνθήκες Είχα την ευκαιρία πριν από λίγα χρόνια να μεταβώ και στο Ισραήλ και στη Λόριδα της Γάζας και είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάς ποτέ. Έχεις την εικόνα αυτή πάντα στα μάτια σου Όταν βλέπεις πώς ζουν εκεί τα παιδιά και πώς μεγαλώνουν, το είπατε κι εσείς, ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ουσιαστικά να φροντίσουμε να ε, επέλθει η απαραίτητη πολιτική λύση ε, στην περιοχή. Κάτι που είδα στο φυλάδιο και δεν αναφερθήκατε, μπαίνοντα πήρα το φυλάδιο αυτό, ε, ισότητα των φύλων. Ε, τι γίνεται με τις γυναίκες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ρωτήσω τι κάνετε ακριβώς για τις γυναίκες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στην Επιτροπή μας. Όποιο έχει πάει σε καταβλισμό προσφύγων καταλαβαίνει τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να ζεις εκεί πέρα και να επιβιώνεις. Σας ευχαριστώ ε, που το αναφέρετε στο φυλάδιό σας, αλλά θα με διέφερε πάρα πολύ να μας πείτε περισσότερο εδώ. Όπως επίσης και το πώς βλέπετε την πολιτική λύση της ε, σύραξης, πώς μπορεί αυτή να Ξέρω ότι αυτό που σας ρωτάω υπερβαίνει κάπως την ε, εντολή σας με τη στενή έννοια, αλλά θα μπορούσατε να δώσετε και το όραμά σας, τη θεώρησή σας για την πολιτική λύση εκεί. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Uh, Ευχαριστώ, πρόεδρε, λέει ο κύριο Σμιθ. Σας ευχαριστούμε, Πιέρ, για τα όσα μα ε, είπατε, που ήρθατε να μα ενημερώσετε. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας, το θυμό σα ακόμη. Πάντως συγχαρητήρια στην οργάνωσή σας και εδώ στο Γραφείο των Βρυξελών που μας ενημερώνετε και οργανωτικά και για τις εξελίξεις της επιτόπου. Έχετε δίκιο που να συνεχιστεί η δέσμευσή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς οι ρίζες του φαινομένου βρίσκονται αλλού, βρίσκονται στην Βρετανική Αυτοκρατορία και εγώ ως Βρετανός και Σκοτσέζος ξέρω ακριβώς τι έγινε και ξέρω τις συνέπειες. Λοιπόν σήμερα είναι ε, η πηγή των παλαιών ε, αδικιών. Ε, μας λέγατε για 5 εκατομμύρια προσφύγων στην Νορβηγία, μα τόσοι είμαστε όλοι όλοι οι Σκοτσέζοι σήμερα, είναι απίστευτη η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τις συνέπειες του ότι πώς η ριζοσπαστικοποίηση η απελπισία. Και τα λέγαμε ακριβώς τα ίδια και με την Συριακή Αντιπολίτευση την εβδομάδα εδώ στις ε, ε, Βρυξέλλες και βέβαια οι συνέπειες θα είναι τρομερές για την περιοχή όλη, για, όλο τον κόσμο. Ε, πρέπει να συνεχιστεί η προσοχή μας, αλλά ε, μιλάμε τώρα για κάποιες συνέπειες οπότε και εσείς θα πρέπει να αρχίσετε να ασχολείστε περισσότερο με τις αιτίες του φαινομένου, με τις αιτίες αυτής της κατάστασης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το Ισραήλ που είναι μια δημοκρατία. Εκεί υπάρχουν δυνάμεις διαλόγου και πρόοδο. Είναι μια κοινωνία περίπλοκη. Είναι δημοκρατία. Η Συρία δεν είναι δημοκρατία. Άρα υπάρχουν ε, φωνές και πρόσωπα ε, στο Ισραήλ που να είναι συνομιλητές μας. Να επομένως μία αφετηρία εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου και δεν θέλω να ευνοήσω καμία πλευρά. Υπάρχουν πάνω από δύο πλευρές στην υπόθεση αυτή. Έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε και δύο παράλληλα σύμπαντα. Έχουμε μια μεριά τη διεθνή κοινότητα που συνομιλεί με το κράτος Ισραήλ αλλά επιτόπου εκεί υπάρχουν οι δυνάμεις που καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε μακρόπνοη λύση. Όπως είπατε και εσείς, ζουν σε άλλους πλανήτες εκεί. Χωριστά τελείως. Και αυτό φυσικά κάνει τον διάλογο. Τελείως αδύνατο και τις διεθνείς προσπάθειες χωρίς νόημα. Γι' αυτό σας είπα, λίγο παραπάνω ούτως το την εντολή σας. Και εσείς είσαστε αντικειμενικός παρατηρητής, αλλά για πέστε μου, από αυτής τη πλευράς, σε ποιον μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα, ποιον να πιέσουμε στο Ισραήλ τόσο ώστε να αρχίσουν κάποιες διαπραγματεύσεις που να έχουν νόημα. Έχουμε ένα σωρό συναντήσεις και επαφές ε, χωρί νόημα, αλλά έχουμε αυτή την αναστολή των συμφωνιών σύνθεσης, σύνδεσης, ε, το, το, μπορεί να πιέσουμε και, με αυτό, μπορεί να πιέσουμε και με το Horizon 2020, μπορέσουμε να πιέσουμε κάποιους στην Ισραηλινή κοινωνία και έτσι επομένω να κάνουν το τραπέζι Ισραηλινή για κάποιες διαπραγματεύσεις με νόημα που να φέρουν τη διαφορά. Καταλαβαίνω γιατί είσαστε απεσιόδοξος. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα λεφτά τα οποία θα προδώσουμε στην Ούδε για να υπάρχει μια λύση πολιτική. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο πάλι. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κ. Καστάλτα. Να ευχαριστήσουμε τον ε, ε, τον Επίτροπο της Σούνρα που τον σημερινό μας προσκεκλημένο για τα όσα ε, μας είπε. Ήταν ε, πάρα πολύ ευγενικό αυτό το οποίο είμαστε οι πρώτοι δωρητές για τον φορέα του. Και ελπίζουμε ότι θα πρέπει να βρούμε τα σχετικά ποσά και ελπίζω να αυξηθούν κιόλα. Άκουσα τι είπε η κυρία Βαλενθιάνο. Και συχνά και εμείς ακούμε επικρίσεις. Επικρίσεις και από άλλους συναδέλφου, αλλά και από την κοινωνία, ότι δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πιάνουν τόπο. Μπάς και καταλήγουν κιόλας και στους εξτρεμιστές. Εσείς, τι έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια για να μπορέσετε να έχετε κάποιες εγγύσεις για το ότι αυτή η χρηματοδότηση δεν πάει αλλού από εκεί που θα έπρεπε. Επίσης, σε σχέση με αυτά που λέγατε προηγουμένως όσον αφορά την έλλειψη προοπτικών για μια ολόκληρη γενιά Παλαιστινίων στην Γάζα. Και ε, αυτό δεν μπορεί να εκπλήξει κανέναν ότι έτσι πιάνουν τόπο η, πιάνει τόπο η, το έργο των εξτρεμιστών Και ακόμα και το ίδιο η ζωή έχει χάσει το νόημά εκεί πέρα. Έχουμε εξέλιξη μέσω αυτής της σύγκρουσης, τώρα έχουμε έναν ε, πόλεμο. Κάποτε ήταν, ε, ήταν ε, ο πόλεμος κατά του κατακτητή από πλευράς του κατακτημένου σε μια κατάσταση κατοχής, τώρα είναι πόλεμος πολιτισμός και θρησκειών. Οπότε να δούμε να δούμε πώς τώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις να ξανανοίξει το αεροδρόμιο της Γάζας, να ξανανοίξει η Γάζα στον κόσμο. Να σταματήσει αυτή η πολιορκία που σοβήκε τόσα χρόνια. Μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς θα βοηθήσουν τον έλεγχο των συνόρων και να υπάρχει από την άλλη μεριά και έγκυση των Παλαιστινίων μπορούν να έχουν χθε την πόρτα στον κόσμο αλλά και από την άλλη μεριά να μπορέσουμε να πλησιώσουμε και τους Ισραηλινούς που θέλουν κάποιο στάνταρ ασφάλειας. Τέλος, μας μίλησατε για την ε, Συρία, για τις τελευταίες αυτές πιο πρόσφατες τραγωδίες που οδήγησαν τόσους σε Λίβανο, σε Τουρκία, σε Ιορδανία Είδαμε όμως ότι όσον αφορά την Τουρκία έχουμε πολλές ε, αντιτιθέμενες φωνές για το τι γίνεται με τους ε, Παλαιστίνους αλλά και Σύριους πρόσφυγες που πάνε εκεί. Γιατί ε, ακριβώς συγγενεύουν ιδεολογικά αυτοί οι πρόσφυγες λένε με κάποιους άλλους εξτρεμιστές που δρούν εκεί στην Τουρκία. Α δούμε επομένω τι θα γίνει και βέβαια δεν μπορούμε παρά να ε, εκτιμήσουμε αυτό το φόρο αίματος που εκπληρώσει η οργάνωσή σας, όπως είπατε. Οπότε για άλλη μια φορά τις, τα θερμότερα συγχαρητήριά μας και ευχαριστήρια μας για το έργο σας. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος, δίνει το λόγο στον επόμενο. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τη φωνή μου δεν είναι αποτέλεσμα ουισκοποσίας αλλά κρυώματος η φωνή μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ επακριβή παρουσίαση της κατάστασης και τα στατιστικά στοιχεία που μας δώσατε. Έχω δύο παρατηρήσεις και δύο ερωτήματα. Αναφερθήκατε στην κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης στην Παλαιστίνη. Εγώ έχω πάει στους τελευταίους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου πέρσι στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Μας είπανε ότι και η Χαμάς είχε επιβάλει αποκλεισμό στην Γάζα σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά υλικά. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει ή όχι. Και επίσης τι σημαίνει πια η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην ε, Παλαιστίνη που υπήρχε στα χαρτιά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει στην πράξη. Επίσης είπατε για τις υποσχέσεις που δόθηκαν στη συνδιάσκεψη της, ε, του Κάιρο. Ποιοι είχαν υποσχεθεί τι και ποιοι δεν τήρησαν τις υποσχέσεις αυτές. Γιατί ίσως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε και κάπου αλλού. Και επίσης αναφέρατε τη σημασία της διπλωματικής ε, προσπάθειας του διαλόγου. Έχουμε μεγάλη δυσκολία να πάμε στη Γάζα, το είπαμε και αυτό όταν πήγε η τελευταία μας αντιπροσωπεία από τους σοσιαλιστές προς τον ε, πρόοδο του Κοινοβουλίου, οι γερμανικοί φορείς, τα ιδρύματα της Γερμανίας μπορούν να μπουν στη Γάζα, αλλά όχι εμείς ως κοινοβουλευτικοί. Βλέπετε να υπάρχει κάποια δυνατότητα να το τροποποιήσουμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε δυνατότητα να είμαστε παρόντες εκεί και να συζητήσουμε με τους συνομιλητές μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος πάλι χωρίς μικρόφωνο βέβαια και δίνει το λόγο ο κ. Σαφχάζων. Ο κ. Σαφχάζων με μικρόφωνο. Τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση Λαμβάνοντας υπόψη ότι διαχειρίζεστε τόσο καλά όλα αυτά τα προγράμματα και δεν θέλω να αμφισβητήσω τις ικανότητές σας γιατί τα αραβικά κράτη δεν συμβάλλουν περισσότερο στο έργο της Ούντρα ε, και μάλλον γιατί δεν συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της περιοχής αυτής και λαμβάνοντας υπόψη το κενό που έχετε στον προπολογισμό σας έχετε ζητήσει περισσότερα κονδύλια από αυτούς και σας έχουν πει ότι θα τα δώσουν ή όχι. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την ερεσιμότητα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια. Πιστεύετε ότι η κύρια μέρημνα της Φατάχ και της Χαμάς είναι η ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία ή είναι η μάχη εναντίον του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Είναι η προτεραιότητά τους η ανάπτυξη και η δημοκρατία ή ο αγώνας κατά του Ισραήλ. Τρίτη παρατήρηση. με κάποιο τρόπο εσείς ουσιαστικά και για διάφορους λόγους υποκαθιστάτε τις τοπικές κυβερνήσεις. Για σας είναι καλό αυτό, το ότι παίζετε το ρόλο των κυβερνήσεων που δεν είναι σε θέση να δράσουν. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα τα οποία ήθελα να σας θέσω και θα ήμουν ευγνώμων να μπορούσατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον καλεσμένο μας, ο κύριος Χάν. Και να σας συγχαρώ και εσάς και τον φορέα σας για το τόσο ικανό έργο που κάνετε σε τόσο δύσκολες συνθήκες, όχι μονάχα με τα με, τα, με τους οικονομικούς περιορισμούς που έχετε, αλλά και τους άλλους περιορισμούς. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Βλέπουμε ότι ο λαός της Παλαιστίνης υποφέρει και η κατάστασή του επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ για το γεγονό που, όπω λέτε, 42% των Ισραηλινών δεν έχουν έρθει ποτέ πρόσωπο, με, ένα Ισραηλ, με ένα Παλαιστίνιο. Ο κόσμο πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα για μια δίκαια και μόνιμη ελ, ελπίδα λύση για του Ισραηλινού και του Παλαιστίνιου στο πλαίσιο ενός καθεστώτος δύο κρατών. Αλλά όταν δεν έχει υπάρξει αυτή η επαφή, 42% δεν έχουν συναντήσει ποτέ κάποιον από την άλλη πλευρά, αυτό τροφοδοτεί το φόβο και την ικανότητα δαιμονοποίησης της άλλης πλευράς. Όλοι μας <clears throat> θέλουμε να δούμε να υπάρξει περισσότερη κινητοποίηση για τα θέματα αυτά. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο για να βοηθήσει την εξέβρεση μια λύσης στην ε, περιοχή. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν απολέσει ένα μέρο τη αξιοπιστία, του είναι φανερό ότι χρειάζονται περισσότεροι οι οποίοι θα εμπλακούν για την αναζώτηση μιας ε, λύσης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, στο φως όλων αυτών των στατιστικών, πόσο σημαντικό θα ήταν να σταματήσει αυτός ο αποκλεισμό ο οποίος στραγγαλίζει τη Γάζα και την κάνει μια ανοιχτή φυλακή. Θα ήθελα επίση να ακούσω από εσά. Τι είδους μέρισμα ειρήνης θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε αν υπήρχε κάποια λύση μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ σε σχέση με τον αγώνα κατά του εξτρεμισμού που βλέπουμε να αναδύεται σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο χωρίς μικρόφωνο πάντα, ως ήθισε. Δίνει το λόγο και πάλι στον καλεσμένο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσει Πρώτα απ' για να ξεκινήσουμε με την κυρία Βαλενθιάνο ε, για το ότι, ότι υποστηρίζουμε το, το σύστημα αυτό ε, και το τι έγινε μετά την διάσκεψη του Καΐρου. Μα είχαμε πάρα πολλές στιγμές όπου πάρα πολλά κράτη που πήγαν στο Γάρο αναρωτήθηκαν μα έχει νόημα τώρα να επενδύουμε χρήματα στη Γάζα μα ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει αυτός ο, ο κύκλος ανασυγκρότησης καταστροφής ε, το τόνισε αυτό και ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επανειλημμένα. Οπότε και εμείς αναρωτηθήκαμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, μπορούμε να συντηρήσουμε την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή όχι. Και εγώ πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι για τις χώρες ε, που οι πρόσωποι τους μου είπαν ότι αντιμετώπισαν αυτό το δίλημα. Οι χώρες εκείνες που ε, δίστασαν να εκτανίσουν χρήματα για την Γάζα. Μα είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα ισχύει. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ακόμα κρατιούνται όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τη Γάζα ακριβώς για τους λόγους αυτούς. Οπότε θα πρέπει να απαντήσω το εξή. Δεν μπορούμε. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κρατιούνται. Δεν μπορούν να συγκρατούνται από το να συμβάλλουν σε ανθρωπιστική ε, βοήθεια και από την Ελλάδα θέλουν ότι ασκούν πολιτική. Συμπαθάτε με, αλλά γίνεται τίποτα άλλο. Αν αποφασίζει μια κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να δώσει χρήματα για τη Γάζα σήμερα, ε, τότε ε, τουλάχιστον κάντε κάτι. Κάντε κάτι στο πολιτικό μέτωπο. Αλλά δεν είναι δυνατόν κανείς να φρενάρει και στο μέτωπο τη οικονομικής ενίσχυση και της πολιτικής. Αλλιώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα προσπαθούσαμε, θα προτιμούσαμε να υπάρχει κάτι για τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τις στοιχειώδεις ανάγκες αλλά το κάνει κανείς ε, ούτε το ένα ούτε το άλλο ε, τότε γυρνάει την πλάτη σε αυτή την τρομερή κατάσταση. Γι' αυτό και τι προέκυψε. Τι επανειλημμένα ελέγχθηκε μετά από την ε, Ποιος εξελίξει εκεί τι ε, λέχθη. Το το τα είπε και η κυρία Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε η Γάζα να συνεχίσει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν, πριν γίνει ε, ο αποκλεισμό. Θα πρέπει τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει από πολιτική πλευρά. Η Ούνρα δεν έχει εντολή να παρεμβαίνει πολιτικά Όμω, όσο εκ της θέσεώς μα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συνέπειες από την έλλειψη πρόοδου στο μέτωπο της πολιτικής λύσης. Να. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Άρα, χρειάζονται πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Από πολλούς, από πολλές πλευρές, αλλά όλη αυτή η αστάθεια που τώρα διαπιστώνεται στην Μέση Ανατολή τελικά έχει γίνει θέμα ευρωπαϊκό επιτρέψτε μου να πω. Γιατί εσείς είσαστε παράγον διατήρησης προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς έχετε ανλάβει να υποστήξετε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλα όσα γίνονται εκεί πέρα είναι η άρνηση της αξιοπρέπειας, αλλά υπάρχει και το θέμα της σταθερότητας. Αυτά λοιπόν μπορούν να συνδυαστούν και θεωρητικά και πρακτικά. Άρα έτσι μπορεί κανείς να ενατενίζει το μέλλον. Ευχαριστώ για τόσα είπατε επίσης όσον αφορά ε, για τις απώλειές μας. Αναγνωρίζετε το τι γίνεται από το προσωπικό μας. Έχουμε 30.000 30.000 προσωπικό δικό μας. Σημαντική παρουσία. Και από τον Ερθό Σταυρό που έχω δουλέψει εκεί, ξέρω δεν υπάρχει κάποιος άλλος με τέτοια επίδοση. Και είπαμε χάσαμε 11 στη Γάζα, 14 στην Συρία και συνεχίζουμε. Οπότε αυτά δεν σας τα λέω για να κομπάσω όσον αφορά αυτά τα νούμερα. Αλλά θα σας πω ότι είναι συνάδελφοι αυτοί, αναλαμβάνουν κινδύνους, άφησαν τις οικογένειές τους. Απογειώνουν την οικογένειά τους το πρωί και δεν ξέρουν αν θα ξαναδούν το βράδυ και πάνε στους καταβλισμούς, στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Εδώ σε αυτό είναι πολύ αξιοπρόσεκτο. Είναι και το θέμα της ισότητας των φίλων, κάτι το οποίο εμείς το έχουμε ως φιλοσοφία από όταν άρχισε να λειτουργεί ο φορέας μας. Ε, κάποιες από τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ έχουν ασχοληθεί με την παιδεία και με άλλες πρωτοβουλίες στο Αφγανιστάν, ας πούμε, και ξέρετε το θέμα της ισότητας και εμείς έτσι λειτουργούμε έχουμε περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές στα σχολεία μας και όλα αυτά τα κάνουμε με αντιμετώπιση ισότητας ισότητας των φίλων αλλά τι γίνεται όταν φεύγουν τα κορίτσια από το σχολείο ε, το πολιτικό περιβάλλον μπορεί να υπονομεύσει τις δυνατότητες αυτών των νέων κορισιών σε σχέση με το αν μπορούν να κάνουν κάποια αστιαδιοδρομία, να γίνουν γιατροί και μηχανικοί και δάσκαλοι όπως βλέπουμε να γίνονται στα σχολεία μας. Επίσης, ρωτήσατε ποια θα μπορούσε να είναι η πολιτική λύση, πώς το βλέπουμε εμείς. Ε, αυτό είναι το όριο της εντολής μας. Δεν μπορούμε εμείς να χαράξουμε αυτή την πολιτική λύση. Αλλά μετά από τόση δουλειά σε τέτοια εκεί μέσα στη σύγκρουση, θα πρέπει να ρωτηθούμε ποιο είναι το κόστος του ΡΥΠΗ επί τόσα χρόνια δεν έχει δοθεί μια λύση. Άρα δεν είναι η ερώτηση ποια είναι η λύση, αλλά ποιο είναι το κόστος απουσίας της λύσης. Τι σκέφτεστε εσείς. Η απουσία πολιτικής λύσης και πολιτικής δέσμευσης σε τι οδήγησε. Δεν οδήγησε σε ριζοσπαστικοποίηση. Σκεφτείτε ένα Παράδειγμα, μια κατάσταση που δεν έλαβε κάποια πολιτική λύση, οπότε και είχαμε ριζοσπαστικοποίηση. Μεγάλο το κόστος του να μην δεσμεύεται κανείς να δοθεί μια λύση. Όπως είπατε, πρόκειται για αγανάκτηση. Γιατί οι πολιτικές προσπάθειες, οι προσπάθειες πολιτικής λύσης είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις κοινότητες. Ναι, προσπαθούμε να προβάλλουμε όσο μπορεί περισσότερο τα πράγματα και στη Γάζα αυτό που κάναμε όσο γίνεται να, να, προβάλλουμε τις θέσεις μας γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν έχει σημασία πόσο καλός είναι κανείς το ανθρωπιστικό έργο και πόσο αποτελεσματικό στο ανεπτυξιακό έργο. Ποτέ καμία βοήθεια δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, ναι, θα πρέπει αυτές τις υπηρεσίες να τις ε, προσφέρουμε, αλλά επίσης θα πρέπει να μην σταματάμε τι σημαίνει για τους πρόσφυγες να μην έχουν δικαιώματα, να μην έχουν αξιοπρέπεια. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε το ποια θα είναι η πολιτική λύση. Αυτό είναι πέρα από τα όρια μας. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται στράτευση, χρειάζεται ανάληψη κινδύνου και εσείς όμως από την άλλη μεριά είσαστε ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ξεπερνιούνται οι επιφυλάξεις, οι σκεπτικιστές. Ξέρω πάρα πολλοί αμφιβάλλουν, είναι απεσιόδοξοι για την Μέση Ανατολή. Αλλά ε, εκεί το να αμφιβάλλει κανείς για, για την ειρήνη είναι κανείς σαν να σηκώνει τα χέρια. Το 1946 1947 πόσοι είχαν επιφυλάξεις για την ειρήνη στην Ευρώπη. Όσοι θα υπήρχαν σε μια αίθουσα που θα έλεγαν ότι ναι, θα υπάρχει ένα μέλλον στην Ευρώπη, κάποια στιγμή θα υπάρχει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Κοινή Θεσμή, θεσμικά όργανα. Σήμερα το θεωρούμε αυτονόητο. Καλά, εγώ είμαι Ελβετό, <laughs> δεν θα έπρεπε να επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά πολλοί εσεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρείτε αυτονόητα όλα αυτά. Και όμω ε, θεμελιώθηκαν, βασίστηκαν και χτίστηκαν σε μια διαιρεμένη Ευρώπη υπό κάθε έννοια διχασμένη. Ε, στη Μέση Ανατολή χρειάζεται πολιτική βούληση και είναι κάλλιστα εφικτό κάτι τέτοιο εάν ε, υπάρξει η βούληση και ε, διοχετευτεί και η απαραίτητη ενέργεια. Και είναι και απαραίτητο και για την περιοχή αυτή και για τον κόσμο ολόκληρο. Ο κύριος Καστάλντο ε, ρώτησε τι εγγύησεις έχουμε για τη χρηματοδότηση και πώς θα πιάνουν ε, τόπο τα λεφτά και θα πηγαίνουν ε, στους δικαιούχους. Στη Γάζα έχουμε προσωπικό 12.500 και μία από τις μεγάλες μας ισχύσεις είναι ότι δεν έχουμε ε, εταίρους που ε, τα εφαρμόζουν και τα ελοποιούν στην πράξη. Είναι ήδη μας υπάλληλοι και έχουμε άμεση επαφή και ίδια ε, γνώση για το τι συμβαίνει επί τόπου. Και αυτό το θεωρώ από τα μεγάλα μας ατού. Να σας πω μια συζήτηση που είχα στο τέλος μετά τη σύραξη στη Γάζα με κάποιον από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και το λέω γιατί είναι κλειδί για μένα και ο διάλογος με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε ισχυρή δέσμευση και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με άλλους και με τι ένοπλε δυνάμει Δεν συμφωνούμε πάντα, προφανέ είναι αυτό, έχουμε τι διαφωνίε μας, αλλά και αυτό ακριβώς είναι τμήμα ενό διαλόγου. Είναι να συμμετέχεις. Αυτό εννοώ ότι έχουμε μπλοκή εκεί και τελικά όταν τελείωσε η σύραξη το ρώτησα. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς που φέρνουμε τσιμέντο στη ε, Γάζα για την ανοικοδόμηση ε, βρέθηκε ποτέ στις σύραγγες και η απάντηση των Ισραηλινών ήταν σαφέστατη. Όχι. Δεν υπήρχαν στοιχεία ότι οποιαδήποτε δομικά υλικά ή άλλα χρησιμοποιούσαμε και μεταφέραμε εκεί, εμείς δεν βρέθηκαν στις σύραγγες. Και παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχει το Ισραήλ μαζί μας για διάφορα θέματα, τα συζητούμε και διαφωνούν και αυτοί με που λέμε και κάνουμε, αλλά έχουν και αναγνώριση για το τι κάνουμε και ε, ελέγχουμε ε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για να μην πέσουν σε λάθος χέρια, όποιοι και να είναι αυτά. Ε, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει ένα θέμα με τη ριζοσπαστικοποίηση τη μελλοντική στην περιοχή. Κοιτάξτε, εκεί ε, ζουν νέοι ε, σε καταβλισμό, στο σε διάφορους καταβλισμούς του Λιβάνου και παντού στη λωρίδα της Γάζας. Ζουν σε καταβλισμούς με πάρα πολύ λίγες προοπτικές για το μέλλον τους και η ριζοσπαστικοποίηση καμιά φορά είναι και ένας πειρασμός γιατί είναι βαθιά ε, οργισμένοι και βαθιά αγανακτισμένοι και η δική μας επένδυση στην παιδεία είναι πραγματικά κλειδί. Γνωρίζετε ότι αυτόν τον καιρό Σύριοι πρόσφυγες δεν έχουν σχολεία. Έχει βρει τρόπο η ΟΥΡΑ επί σειρά δεκαετιών να φέρνει στο επίκεντρο των προσπαθειών της ε, τα σχολεία για να μπορούν οι νέοι, τα παιδιά να αποκτήσουν ε, ιδιότητες, δεξιότητες, να μορφωθούν, να έχουν ένα μέλλον με προοπτικές. Αυτό είναι μια επένδυση που πιάνει τόπο και εσείς μας δίνετε τα μέσα για να το κάνουμε. Θα χρειαστούμε περισσότερους πόρους, αλλά ήδη μας τους δίνετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της περιοχής. Ωστόσο, και θέλω να το τονίσω αυτό και πάλι, εάν τα παιδιά που πάνε στα σχολεία μας βγαίνουν και δεν έχουν καμία προοπτική να εργαστούν τελικά, τότε η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Αυτό έχει να κάνει όμως περισσότερο με την κατοχή και τον αποκλεισμό της ζώης της Γάζας. Και εγώ επικεντρώνομαι πάρα πολύ στα δικαιώματα των ε, Παλαιστινίων προσφύγων, γενικότερα τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ε, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αυτό είναι ένα ε, γνώμονας για μας. Κύριε Λίτς, ε, μιλήσατε για τον αποκλεισμό και το ρόλο της Χαμάς στην ανοικοδόμηση. Είναι γεγονός και σαφές ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενέχονται εκεί ε, για την καθυστέρηση της ανοικοδόμησης από τότε που ήταν η τελευταία σύρεξη. Το ένα είναι το κυβερνητικό κενό. Δεν υπάρχει στενή συνεργασία που χρειάζεται ε, μεταξύ των αρμοδίων κρατικών αρχών ε, στη Ραμάλα, την ε, κυβέρνηση Εθνική Συνένεση και ε, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χαμάς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι θέμα αυτό. Και ένα άλλο θέμα είναι και η χρηματοδότηση. Και ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για την εισαγωγή δομικών υλικών ξεκίνησε αργά, αλλά τώρα επιταχύνει. Ελπίζουμε να επιτεθεί κάποια πρόοδος εκεί, αλλά είναι ευαίσθητα τα πράγματα. Για το Κάιρο ζητήσατε στοιχεία και αριθμητικά στη διάσκεψη του Καϊρού εμείς για την ανοικοδόμηση και για τις επισκευές ε, και τις επιδοτήσεις ε, ε, των ανοικίων ήταν 720 ε, εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έχουμε 175 εκατομμύρια υποσχέσεις. 125 είναι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και 100 έχουν ήδη δαπανηθεί. Όσα είχαμε για την ανοικοδόμηση των ε, οικειών. Όσα είχαμε. Έχουν ήδη ε, εκτεμιευθεί Ευτυχώς Πρόσφατα είχαμε και νέες δεροές αλλά παραμένει μεγάλο το χάσμα. Από τα 720 που είχαν υποσχεθεί, 175 έχουν έρθει μόνο. Θα πρέπει λοιπόν όλε οι χώρε που έδωσαν αυτέ τι υποσχέσει στο Κάιρο και δεσμεύτηκαν θα πρέπει τώρα να τι υλοποιήσουν. Και εμεί δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε το μέρο που μα αναλογεί. Ε, πόσο δύσκολο οι βουλευτέ να μεταβαίνουν και Το άκουσα κι εγώ αυτό, ναι. Εμεί μπορεί να μην έχουμε τη λύση για να σας ανοίξουμε την πόρτα να μπείτε, αλλά αν έρθετε μπορούμε να διευκολύνουμε επιτόπου τις επισκέψεις και γίνονται πολλές επισκέψεις για οι υπουργοί και βεβαίως η κυρία Μογκερίνη όπως σας είπα. Προσωπικά πιστεύω ότι τίποτα ε, δεν είναι ε, καλύτερο από το να πάτε επιτόπου να δείτε εσείς όμως και να ε, μιλήσετε και, και στη Γάζα και στη Βαλαιστίνη, στη Δικαιόχτη δηλαδή και άλλο. Με ρωτήσατε για τις συνεισφορές στην ούνζα Μια στιγμή να το βρω. Α, οι Αραβικέ χώρες, ρώτησε ο κύριο Σαφάουζερ. Αν κοιτάξετε γενικά τη δαπάνη, 1,2-1,3 δις, ο πρώτος μεγαλύτερος δωρητής παραμένουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, δεύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά μια σειρά άλλων κρατών, μεταξύ αυτών και η Ιαπωνία. Ο τρίτος μεγαλύτερος δωρητής μέχρι τώρα είναι η Σαουδική Αραβία και, και τα Εμμυράτα ε, είναι η έβδομη. Ε, ε, οι, χώρες, οι αραβικές χώρες του κόλπου πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα, ακούγεται αυτό, συμβαίνει ήδη. Δεν είναι στον πλήρη βαθμό οι ποσόν που έχουν δεσμευτεί να δώσουν. Ιδιαίτερα, μιλώ για τον τακτικό μας προϋπολογισμό, έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν περισσότερο. Αλλά ε, τρίτος ζωητής σήμερα είναι η Σαδική Αραβία, θα πρέπει να τονιστεί αυτό και να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, ρωτήσατε κάτι άλλο για την αιρεσιμότητα. Η Φατάχ και οι Χαμάς τι στόχο έχουν, την ανάπτυξη ή το ε, πάλι κατά του Ισραήλ. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολιτικό θέμα. Μπορούμε να έχουμε συζητήσεις με ποικίλε γνώμες και απόψεις. Είναι σαφές ότι όταν ο πληθυσμό είναι υποκατοχή εκεί, περίπου 50 χρόνια τώρα, το θέμα των σχέσεων με την κατοχή και με την ε, κατάσταση εκεί επηρεάζει πάρα πολύ τώρα. Κατά πόσο επηρεάζει τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς επιτόπου, δεν θα μιλήσω εγώ εξ ονόματός τους. Αλλά από την ευρωπαϊκή σκοπιά όλοι καταλαβαίνουμε σε μεγάλο βαθμό τι σήμαινε η ε, σύσταση του κράτους του Ισραήλ, τι σήμαινε η ανάγκη των Ισραηλινών πολιτών να αισθάνονται ασφάλεια και ε, στην περιοχή και σε σχέση με τους γειτονές του. Καταλαβαίνουμε αυτό ε, τι σημασία έχει και δεδομένης και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όχι μόνο το δικαίωμα στην ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά και το δικαίωμα να ζει ε, ε, σε συνθήκες ασφάλειας. Αλλά αυτό αν σημαίνει ότι είναι εις βάρος μιας ολόκληρης άλλης κοινωνίας και τις δυνατότητες, την επιβίωση και την αξιοπρέπειά τους και τη δυνατότητα να χτίσουν το ίδιο τους το μέλλον, είναι κάτι το οποίο έχει επιπτώσει σε ανθρώπινο επίπεδο μια ολόκληρης κοινωνίας. Ρωτήσατε για την υποκατάσταση ε, των κρατικών θεσμών. Να σας πω το εξής. Όταν ε, συστήθηκε η Ούνρα, δημιουργήθηκε για να προσφέρει βοήθεια και ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες τα πρώτα λίγα έτη. Διότι η ιδέα ήταν ότι θα βρεθεί μια λύση και ο κόσμος θα γυρίσει στις αιστείες του και θα καταργηθεί πολύ γρήγορα η ώρα γιατί δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Πράγμα που δεν συνέβη. Ε, τα, οι σημαντικές εξελίξεις ήταν όταν κατάλαβε η ΟΥΝΡΑ και τα κράτη το υποστήριξαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι ένα τμήμα της εντολής μας θα το μετατοπίσουμε για να παρέχουμε και υπηρεσίες. Όχι απλώς ανθρωπιστική βοήθεια, ε, αλλά να επενδύσουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι τεράστια επένδυση, βασική για την περιφέρεια και για τη μελλοντική της σταθερότητα. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει σχολείο, έχουν εμορφωθεί έχουν ικανότητες, δεξιότητες για το οποιοδήποτε μέλλον της περιοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν εμείς δεν υποκαθιστούμε κρατικούς θεσμούς, διότι τα κράτη στην περιοχή δεν είναι έτοιμα τώρα να αναλάβουν ε, τα όσα εμείς παρέχουμε στους πρόσφυγες. Ούτε οι Λιβανέζοι μπορούν, γιατί εμείς είχαμε αυτό το ρόλο, ούτε στην Ιορδανία. Έχουν πολλή δουλειά οι Ιορδανοί τώρα ήδη ε, με τους Σύρους πρόσφυγες. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο είναι τι σημαίνει να έχουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει εκτός από τους Παλαιστίνους πρόσφυγες τώρα ένας δεύτερος παράγων μόνιμης προσφυγιάς που είναι οι Σύριοι πρόσφυγες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ήταν η Ελβετία Λίβανος θα είχαμε τώρα στο μεταξύ 3 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Αυτό ζει ο Λίβανος αυτή τη στιγμή από ποσοστά. Στην Ελβετία Γίνονται πολύ συναισθηματικές ε, φορτισμένες συζητήσεις όταν πρόκειται για 500 ε, πρόσφυγες ε, να φτάνουν και σε άλλες χώρες. Στο Λίβανο έχουν 1,5 εκατομμύριο για να καταλάβουμε και την τάξη μεγέθους και τι περιμένουμε από την Ούρα να κάνει και σε ό,τι αφορά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τις δεσμεύσεις. Και ένα τελευταίο, κύριε Χάν. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που είπα προηγουμένως... Α, ρωτήσατε αν υπάρχουν στοιχεία ότι αν πολιτικά λυθεί αυτή η κατάσταση θα έχει επιπτώσει και σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό. Αλλά πρέπει να πω ότι επειδή έχω εργαστεί σε εμπόλεμες περιοχές στη Νότια Ασία, στη Μέση Ανατολή επί σειρά ετών, σίγουρα το θέμα των ανεπίλητων ε, ζητημάτων του Παλαιστινιακού είναι στην καρδιά πολλών αντιλήψεων και πολλών αφηγήσεων αν ε, είμαστε, είναι η διεθνή κοινότητα ε, δίκαιη και έχει ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση. Το κόστος της ε, παραμέλησης του μέλλοντος Παλαιστίνης είναι πάρα πολύ υψηλό. Και θα σας πω τελειώνοντας αυτή την εντύπωση. Οι Παλαιστίνοι, οι πρόσφυγες που έφυγαν από το Γιαρμούκ, μου είπαν ότι όταν ε, το μέτωπο έφτανε στο Γιαρμούκ, ε, ζούσαν δίπλα σε Σύρους και είπαν ότι εμείς ως Παλαιστινοί αμέσως καταλάβαμε τι γινότανε και τι ερχότανε. Οι Σύροι χρειάστηκαν λίγο παραπάνω για να το καταλάβουν, γιατί ήδη στην ιστορία μας είχαμε ζήσει τι σημαίνει να χάνεις τις αιστείες σου, να χάνεις όλο σου το βιός και ε, το Χόμς στη Συρία που υπάρχει παλαιστινιακός καταβλισμός είδα πως ο, ο κόσμος επιζούσε δίπλα στον Μπαμ Άμερ που καταστράφηκε από τις ε, εχθροπραξίες. Και εξεπλάγει πώς κατάφεραν να επιβιώσουν οι Παλαιστίνοι στον καταβλισμό και μετά κατάλαβα γιατί αν, αν ως Παλαιστίνιος απεμπολίσεις ε, την εστίαση, ε, έστω και αν είναι καταβλισμός το μέρος που μένεις θα το, το κάνεις για πάντα και ο, ο κόσμος πραγματικά αγκιστρώνεται εκεί και θα πρέπει να το δούμε αυτό το κόστος, θα είναι κόστος και σε ανθρώπινους όρους και γενικότερα και στο δωμό της ειρήνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να ζητήσω την κυρία Βαλενσιάνο να αναλάβει την Προεδρία. You speak in Italian, fantastic. Tras la presentación, sí. es el señor que va a hablar. Sí. Primero, que tendría que hablar. Bueno, muchas gracias, colegas. Vamos a... Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε την ημερησία διάταξη. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της έκθεσης του κυρίου Πιγιό, μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα θέματα των προκλήσεων ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και τις προοπτικές πολιτικής σταθερότητας. Σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης θα μας παρουσιάσει ο κύριος Αρτούρο Μπαρέλη, ο οποίος είναι ε, κύριος ερευνητής για τα θέματα αυτά και θα μας δώσει τα φώτα του για την έκθεση του κυρίου Πεγιό και εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα από τα θέματα τα είναι πιο σημαντικά που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια σε όλη αυτή την περιοχή της Μεσάντολης και της Βόρειας Αφρικής την ανάγκη να έχουμε μια κοινή στρατηγική μια στρατηγική πολύπλοκη που πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτή τη στρατηγική δεν, δεν μπορούμε να έχουμε εκεί απλοποίησεις το θέμα του πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τον ε, εξτρεμισμό, τον τζιχαδισμό που καταστρέφει τον αραβικό κόσμο και είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρτούρο Βαρβέλη, ο, ο οποίος είναι ανώτερος ερευνητής στο ΙΣΠΙ στην Ιταλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσατε να λάβω το λόγο. Θα μιλήσω όμως Ιταλικά. Ο στόχος της έρευνας που έχουμε αναλάβει στο ΕΣΜΗ μαζί με τον συνάδελφο είναι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και τελικά να μπορέσουμε να κάνουμε μια καταγραφή της επέκτασης του Ισλαμικού κράτους στο Μαγρέμ και στο Μασρέκ. Δηλαδή πρόκειται για ζώνη που ε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Αλγερία και την Ισία. Ιδίω αυτές οι χώρες και μερικές από αυτές στο μεταξύ όσο εμείς ε, δηλαδή συντάσαμε αυτήν την ε, έκθεση οι χώρες αυτές λέγω υπέστησαν σειρά επιθέσεων από το Ισλαμικό κράτος και επομένως βρίσκονται στο στόχο του Ισλαμικού κράτους στο στόχαστρο. Και επίσης αυτό το οποίο προσθέσει ενδιαφέρον και το οποίο το λάβαμε υπόψη για τη σύνταξη της έκθεσης είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ισλαμικού κράτους, τη ΝΤΑΕΣ και της Αλκάιντα από την άλλη μεριά. Είναι κάποιο είδου ανταγωνιστική συνύπαρξη τη σήμερα ημέρα που βεβαίως αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για την Δύση. Η Αλκάιντα φυσικά παραμένει η ιδεολογική αναφορά και για το Ισλαμικό κράτος. Άρα σε ιδεολογικό επίπεδο δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και επομένως αυτή η πρωτοπορία η ιδεολογική παραμένει. Παρά το ότι ο τώρα δεν έχει το χάρισμα του Μπιν Λάντεν. Έχουμε την ανάδεση λοιπόν του Ισλαμικού κράτους, το οποίο καταρχήν χαρακτηρίζεται από κάτι σαν βασικό, χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή επιζητεί την ίδρυση κράτους. Δηλαδή να υπάρχει κάποια εδαφική επικράτεια. Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι έτσι. Διότι αυτό έχει διαμορφώσει την στρατηγική σε επικοινωνία και σε κατακτήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και για την κατοπολέμηση της τρομοκρατίας. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. που τους διαχωρίζει από την Αλγάιντα είναι η εκτεταμένη χρήση προπαγάνδας. ένα και περισσότερο σε σχέση με το τι έκανε στο παρελθόν η Αλκάιντα με εκείνα τα μηνύματα του Μπιν Λάντεν που τα έστελνε από μια σπηλιά στο Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Επομένω, αυτή η χρήση τη προπαγάνδας η εντατική είναι κάτι το κλασικό από πλευρά ενό αυταρχικού κράτου. Πρώτη φορά τώρα έχουμε ένα τέτοιο ζωοστικό κράτο, αλλά για τη Δύση αυτό είναι γνωστό φαινόμενο. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Με αυτή την προπαγάνδα λοιπόν έχουμε τους εξή δύο στόχους. όσον αφορά σαν Δύση, σαν τον υπόλοιπο κόσμο, να μας τρομοκρατήσουν. Γιατί παραμένουν τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι η ΝΤΑΕΣ. Όμως υπάρχει και μια εσωτερική ούτως λειτουργία. Να υπάρξει δηλαδή μια επικράτεια να την ελέγξουν και επομένως από εκεί να ξεκινήσει αυτή η βίαιη προπαγάνδα που γίνεται όλο ένα και πιο βίαιη. Και με διάφορα μέσα θέλουν να προβάλλουν προς τα την ισχύ τους. Και κάνουν ότι είναι και πιο ισχυρή από την συμπαγματικότητα. Οπότε, είπαμε, πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουν υπό τον τους μια εδαφική επικράτεια. Άλλος παράγον τώρα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη χρηματοδότησή τους. Αυτό έχει ζητηθεί αρκετά στο παρελθόν και έχουμε ένα σωρό φήμες σχετικά για το ποιοι είναι οι χρηματοδότηση απ' έξω που τους δίνουν χρήματα. Ε, τώρα πια αυτό είναι μάλλον ε, περιθωριακή σημασία γιατί η χρηματοδότησή τους βασικά γίνεται απ' έξω αλλά είναι το θέμα τώρα του της εδαφικής κυριαρχίας το πετρέλαιο, η πρόσβαση στο νερό, γιατί υπάρχουν εκεί περιτροπηλικές 40.000 βαρελιών την ημέρα. Ε, αυτό δεν είναι βέβαια καμία τρομερή ποσότητα, αλλά αποτελεί δυνατότητα χρηματοδότηση για τις δραστηριότητε τους. Οπότε το πουλούν και να επομένω πώ ε, μπλέκονται έμεσα διάφορες χώρες. Γιατί και οι Σύριοι και οι Τούρκοι αγοράζουν από αυτό το πετρέλαιο. Να το θυμόμαστε αυτό. και έχουμε και την Κεντρική Τράπεζα της Μοσούλης που προβαίνει σε αυτές τις συναλλαγές. Επίσης έχουμε και τους φόρους που επιβάλλονται Κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό κράτος. Φορολογούν βεβαίω τα περισσοκά στοιχεία των χριστιανών εκεί. Είπαμε ότι είχαμε χρηματοδότηση από Τουρκία, από Ιορδανία, από τα κράτη του κόλπου, έτσι στήσαν το κράτος. Υπήρχε αυτή η γνωστή αμφίβολη ε, σχέση με την ε, Τουρκία. Δεν δώσαν απευθείας λεφτά, αλλά ε, λόγω του κουρδικού ζητήματος υπήρχαν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των δύο. Και έπρεπε η Τουρκία να δει πώς θα διαχειριστεί από μια τους Κούρδους από την άλλη το Ισλαμικό κράτος. Και γι' αυτό και η Τουρκία δεν έχει πλήξει ιδιαίτερα το Ισλαμικό κράτος. Στην αρχή και τα κράτη του κόλφου τους ενθάρρυναν και έμεσα τους χρηματοδότησαν ούτως ώστε να χτυπήσουν τον Ασάντα. Για να δούμε για αυτές τις ε, χώρες μία-μία ανάλογα με το πόσο κίνδυνο διατρέχουν για ε, ε, χάσουν την σταθεροτά τους αυτές οι χώρες. Πρώτα-πρώτα η Ιορδανία. Για πολλού λόγου θεωρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό κίνδυνο για μια τέτοια χώρα, έστω και αν είναι μια χώρα σταθερή όπω η Ιορδανία. Ακριβώ λόγω του πόσο κοντά είναι. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Αλλά γι' αυτό γιατί υπάρχει και εσωτερική απειλή για τη χώρα εκείνη που θα μπορούσε να ε, ξεπηδήσει, ε, όπω τα είπε και ο προηγούμενο ε, ομιλητή. Ακούτε κάτι εκτό μικροφόρου. Παρακαλώ, λέει πρόεδρο, παρακαλώ συνάδελφοι. Έχουμε επομένω την εξάπλωση αυτών των ριζοσπαστικών ομάδων ε, και ότι τώρα μπορούν και στατολογούν μέσα από την Ιορδανία ε, γιατί υπάρχουν ένα σωρό πρόσφυγες εκεί από Συρία, ε, από Ιράκ, από Παλαιστίνη. Εκεί πέρα φυσικά υπάρχει έφορα για τον ριζοσπαστισμό. Οπότε να, έχουμε και αυτούς όλους τους τζιχαντιστές αυτού του ξένου μαχητέ που του λέμε που δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για τι ευρωπαϊκέ χώρες αλλά και για τι Αραβικές και για την ε, Ιορδανία. Ε, Επίση υπάρχουν και διαφορέ μεταξύ διαφορετικών φυλών και επομένω κάποιε αυτέ τι φυλέ για να αντιπολιτευτούν, να χτυπήσουν το Ιορδανικό κράτο, συμμάχισαν με του Ισλαμιτέ και βλέπουμε πώ έγινε αυτή η ταχεία άνοδος του Ισλαμικού κράτου, γιατί Ε, προσπάθησαν να κάνουν κάποιες ε, ε, συμμαχίες με διάφορες φυλές σε Συρία και Ιράκ. Όμως έχουν αντικατασκοπία, επίσης πληροφοριών στην Ιορδανία και στρατό καλά οργανωμένο. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα κίνδυνος, αλλά αν δούμε τώρα που, υπάρχει μικρότερος, α πούμε στο, στο Λίβανο. Στο Λίβανο υπάρχει ε, σεκταρισμός, υπάρχουν διάφορε φατρίες, υπάρχουν εσωτερικέ ε, ε, ισορροπίες, οι οποίες είναι μάλλον πάρα πολύ ευάλωτες και βασικά ποιο είναι το ο τρόπος ανάσχεσης για την επικράτηση του Ισλαμισμού στον Λίβανο. Ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους Ισλαμισμός εκεί που μπορεί να τους ανασχέσει. Δηλαδή είναι η Χεσμολάφ η οποία άμεσα συμμετέχει στον ε, πόλεμο της Συρίας υπέρ του Άσαντ. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Έτσι η Χεσμολάκ μπόρεσε να συγκρατήσει τους Σουνίτες και από την άλλη μεριά όμως προκάλεσε ε, ριζοσπαστικισμό. Κάτι το οποίο σοβεί στην ε, ε, Σουνιτική κοινότητα στον Λίβανο. Υπάρχει και η Νούσρα που είναι μια άλλη παράταξη που είναι κοντά στην Αλκάιντα και υπαγωμένως ότι έχουμε την επέκταση, την, την παρέμβαση του Ισλαμικού κράτου στο Λίβανο και εκεί βρέθηκαν κάποιοι που προσχώρησαν Είπαμε για δημιουργία Ισλαμικού κράτου στον ε, Λίβανο, κάτι το οποίο προέκυψε τον Ιανουάριο 2014 που είχαμε ε, διάφορες συγκρούσεις σε πολλές ε, πόλεις και θερμοκρατικές ενέργειες. μεταξύ Ισλαμιστών και του τακτικού στρατού στον Λίβανο. Έχουμε το θέμα εκεί των το θέμα των προσφύγων των ε, Σύρων και το 2015 σύμφωνα με τον ε, ΟΗΕ θα φτάσουν τους 1,3 εκατομμύρια οι πρόσφυγες των Λίβανο. Πολύ ανησυχητικό. Όπως είπαμε επομένως αποτελεί φραγμό στη Ισλαμικό κράτο η Χεσμολά. Από την άλλη μεριά Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν οι απειλέ διότι ακριβώς η χώρα είναι κατετμημένη. Αυτό παραμένει πρόβλημα. Και βέβαια δεν βοηθάει στην κατάθμιση της χώρας ο πόλεμος στη Συρία. Την Ισία τώρα και Αλγερία. Δύο από τις χώρες με εντοπίζουν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την επέκταση των Ισλαμιστών στη Βόρεια Αφρική. Έχουμε εδώ νέες ε, συμμαχίες, νέες συμπαρατάξεις, αλλά ακόμα και διασπάσεις σε υπάρχουσες οργανώσεις, όπως η, η Αλκάιντα, η Αλκάιντα του Ισλαμικού Μακρέμ. και άλλα σήμη και, και άλλες ομάδες που υπάρχουν που συμμάχησαν με το Χαλιφάτο πέρσι. και στράφησαν κατά της ε, Αλκάιντα κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αυτό ήταν κάποιο είδους ε, ανταγωνισμός, αναμέτρηση στα εσωτερικά ε, αυτού του χώρου του, του του Ισλάμ. Οπότε κάποιες ομάδες δήλωσαν ότι είναι πιστές στην Αλκάιντα αλλά από την άλλη μεριά θεώρησαν ότι, είναι πιο κοντά στο χαλιφάτος νέο σημείο έτσι λοιπόν έγινε η δίσδυση του Χαλιφάτου σε αυτές τις χώρες και ιδίω και στην την εκεί που έχουμε υπανάπτυξη, περιθωριοποίηση πολιτική, έχουμε ε, διάφορους θύλακες ε, εκεί μπόρεσε να πιάσει τόπο το Χαλιφάτο. Βεβαίω υπήρξαν κάποια μέτρα και ο Πρωθυπουργό τη ε, Τινησία ε, έφτιαξε μια τρομοκρατική υπηρεσία η οποία και εξειδικεύτηκε να καταπολεμήσει αυτού του τρομοκράτε αυτές τις ομάδες που όπως είπαμε η ε, που συμμάχησαν με το Χαλιφάτο και έχουμε επομένω περίπου 3.000 τινήσιους που έχουν πάει να πολεμήσουν από τις τάξεις της Αλκάιντα στο ε, Ιράκ. Είναι ανάλογα με το μέγεθος της ε, χώρας ο μεγαλύτερος στρατός ξέρων μαχητών που έχουν πάει στα Συρία και Ιράκ. Και φέτος θεωρείται ότι θα πάνε και άλλοι έχουν αρχίσει να πηγαίνουν, κάτι το οποίο φυσικά αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της χώρας. Λιβύη, τέλος, η χώρα που σήμερα είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από όλες από το Ισλαμικό κράτος το οποίο τώρα δρά στην ίδια τη επικράτεια. Δεν είχε σταθερότητα η Λιβύη, ε, Ο κράτος το οποίο συνέχεια ε, κατρακυλάει προς την ε, αναρχία, δεν μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει όλη τη χώρα, υπάρχουν διάφορες φατρίες που ανταγωνίζονται και συμμαχεί μία κατά της άλλης, αλλά δεν μπορεί καμία να επικρατήσει, καμία από αυτούς να αποτελεί πολιτική λύση. Αυτό επόμενος δεν είναι θέμα των τελευταίων ε, εβδομάδων. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την πτώση του Καντάφη. Έχει καταντήσει λοιπόν η χώρα ε, κάτι σαν καταφύγιο για τους τζιχαντιστές και για την ε, αλκαΐδα του Ισλαμικού Μαγρέμπ. Πρόκειται για διάφορες άλλες πολιτι... ομάδες που κινούνται σαν δορυφόροι τοπικές και είπαμε ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός τζιχαντιστών στη χώρα. Έχουμε κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μιλάμε για χίλιους, δύο χιλιάδες. 800 έλεγε το CNN σύμφωνα με κάποιο ρεπορτάζ δεν νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο, Αλλά οπωσδήποτε σε μια χώρα όπου πρετανεύει η αναρχία όπως τη Λιβύη ακόμα και αυτά τα περιορισμένα νούμερα τζιγαντιστών είναι πηγή προβλημάτων για τη σταθερότητα της χώρας, είναι μια απειλή για την Ευρώπη. Ξεκίνησε το πρόβλημα στην ε, Λιβύη, από αυτούς τους τσιγαντιστές που επέστρεψαν. Πρώτο για ένα εξαρτητικό σώμα το οποίο ε, πολέμησε σε Συρία και Ιράκ. Ε, αφορούσε αυτό το εξαρτητικό σώμα 300. Τάγμα, ας το πούμε. Και αυτοί ε, συμπαρατάχθηκαν και με άλλες ομάδες και έτσι αποτέλεσε ένα Ισλαμικό φύλακα. Το τι έγινε μετά μας δείχνει το τι έγινε όταν ο Χαλίφης, ο Αλμπαγδάτ, αποφάσισε να μπει στη χώρα. Έστειλε κάποιους απεσταλμένους. Για να χαραχτεί η στρατηγική της δίσδυση στη χώρα. Και είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες τι έγινε στη Σύρτη. Πολύ ανησυχητικό. Οπότε και θεωρούμε ότι υπάρχει σχέδιο από πλευράς των τζιχαντιστών. Δεν δρούν τυχαία. Είδατε τι έγινε στη ε, Σύρτη. Στη Σύρτη είναι η γενέτρια του Γκαντάφη. Πολύ ανησυχητικό το ότι εκεί γίνονται όλα αυτά τη βλέπουμε ότι η φυλή που ε, βρίσκεται εκεί, η φυλή του Καντάφη, κατά κάποιο τρόπο ανέχεται ή υποστηρίζει το Ισλαμικό κράτος στη Λιβύη. Πολύ ανισχυτικό αυτό, γιατί πρόκειται για μηχανισμούς που είναι πρωτοφανείς. Οι Σουνίτες επομένως ε, υποστήριξαν πρώτα πρώτα την Αλκάντε τώρα και κατόπιν την ε, ε, το Ισλαμικό κράτος για να πιέσουν τους ΣΥΙΤΕΣ. Όμως δεν είναι οι πρώτοι φανατικοί παρίσταντες στη Λιβύη οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχουν και άλλοι που δρούν εκεί και επίσης μας ανησυχούν και αυτά παίρνουν στα ψηλά των εθνικών. Δεν είναι καθόλου. Η Ανσάλα Σαρία είναι μια ντόπια ομάδα τζιχαντιστών. Αριθμούν τους 10.000 περισσότεροι σε σχέση με τους Ισλαμιστές της Λιβύης. Αυτοί λοιπόν είναι οι ντόπιοι Ισλαμιστές έχουν στρατηγική. Συμμαχίες ε, διαφορετικής γεωμετρίας. Οπότε η Αλκάιντα προσπαθούσε να τους ε, προσετεριστεί. Και σε ε, περίπτωση σύγκρουσης με την ΔΑΕΣ τα πράγματα είναι σχετικά. Γιατί αν γίνει κάποιο είδου διεθνής παρέμβαση, τότε αυτοί οι ντόπιοι τζιχαντιστές φυσικά και θα αντιταχθούν σε αυτή την από το τα έξω ε, παρέμβαση. Και αυτό είναι ενισχυτό επίσης και για τις όμορες χώρες όπως για την Αίγυπτο. Έχουμε τις δυνάμεις του Τομπρούκ, του στρατηγού εκεί που υποστηρίζεται από το εξωτερικό. Έτσι θα δράσουν επομένω οι τζιχαντιστές αυτές τις πόλεις. Αυτά στον μας ε, γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι έχει τα μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναχαιτήσει την, ε, ε, το κοινωνικό κράτος. Τη διαχείριση των συνόρων, την ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση, τις διοκτικές αρχές, όλα αυτά όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το καινούργιο πλαίσιο Κάτι το οποίο συνταράσσει τα θεμέλια του Ισλαμικού κράτους. Είναι το θέμα της μη περιθωριοποίησης της πολιτικής. Γιατί έτσι έγινε. Έγινε περιθωριοποίηση στο Ιράκ. Οπότε και υπήρξε έφορο για να γεννηθούν αυτές οι ακραίες λαμικές ομάδες γιατί στηρίχτηκαν σε κάποιες πολιτικές ομάδες που, που, αισθανόντουσαν ότι δεν εκπροσωπούνται, έχουν μείνει απ' έξω. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και οικονομικά μέσα, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακριβώς εκεί που είναι οι πιο περιθωριοποιημένοι, όπως είπαμε για την ε, Ιορδανία, για την Ισία, για την Αλγερία. Εκεί στα όπλα των προσφύγων, στου καταβλισμού του. γιατί ε, ακόμη μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίε αποτελεσματικέ σε στον τομέα της σταθεροποίησης και της ανάπτυξη Ευρώπη. Και αυτό να είναι το αντιστάθμισμα στον, ε, στο Ισλαμικό κράτος και στην ε, τρομοκρατία. Και αυτές οι πολιτικές ανάπτυξη και σταθεροποίησης της χώρας να χρησιμοποιούνται συνδεσμό η μία προς την άλλη. Όμως, να μην ξεχνούμε τον παράγοντα χώρες του κόλπου. Εκείνες ήταν οι πρώτες χώρες που βοήθησαν και που χρηματοδότησαν και που ακόμη ασκούν πολιτική επιρροή. Για να δούμε τώρα τι άλλους μηχανισμούς έχουμε που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και οι οποίοι τώρα εδώ έχουν σημασία και πρόκειται για τους μηχανισμούς που αποτελούν αντίσταση στις προπαγάνδες της Ευρώπης και έχουμε τώρα αυτά τα προγράμματα τα προγράμματα για τις, για κοινότητε κοινότητες στην Ευρώπη έχουμε τους φόρες Οι ξένοι μαχητές θα παραμείνουν ένα πρόβλημα ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ευρώπη και επίσης έχουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες έχουν υποστηριχθεί μονάχα από μερικές χώρες σε εθνικό επίπεδο. Οι πολιτικές απορριζοσπαστικοποίησης, υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν ατομικά άτομα τα οποία έχουν προσεγγίσει μια ε, ριζοσπαστική Ισλαμική ιδεολογία, αλλά τα οποία μπορούν να ανανύψουν. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, έχουμε πολύ λίγο χρόνο για όλη αυτή τη συζήτηση που πρέπει να λάβει το ε, πρέπει να λάβει χώρα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πεγιόν, ο οποίο είναι και εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <coughs> Καθηγητά, δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Έχετε εστιάσει περισσότερο στι τρομοκρατικέ ομάδε. <coughs> Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει όμως περισσότερο είναι η γενική σταθεροποίηση. Υπάρχουν πολλέ δυσκολίες. Το αν έλεγε κάποιος που από 3-4 χρόνια το πρόβλημα μας είναι το Ισλαμικό κράτος και όχι οι δικτάτορες στην περιοχή αυτή, θα μας εξέπλητε τελείως να το έλεγε κάποιος. Έχουμε ακολουθήσει λοιπόν μια στρατηγική που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά τα τρέχοντα γεγονότα. <clears throat> Αναρωτιέμαι αν εμείς τώρα εστιάσουμε μόνο στην τρομοκρατία, αν πράγματι κάνουμε την προβληματική που θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα βαθιά αίτια που μας έχουν φέρει στην τωρινή κατάσταση. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα τωρινά γεγονότα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις εξέλιξεις. Δηλαδή, μπορεί να λύσουμε το πρόβλημα σε μια χώρα, μπορεί να έρθει σε ένα άλλο μέρος. Έχουμε τώρα πολλούς οι οποίοι έχουν γίνει εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά, αλλά θέλω να σταθώ περισσότερο στην προβληματική που μας νοιάζει περισσότερο εμάς. Λέτε κάτι το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικά ευπρεπές. Λέτε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μία ανισομέρεια, ακόμα και μία σχιζοφρένεια. Υπάρχει μια μονομανία που μπορεί να είναι δικαιολογημένη για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την άλλη πλευρά μια πολιτική διαφορετική. Μπορούμε να μαστιγώνουμε τους ε, ε, συμμάχους μας, αλλά συγχρόνως δεν έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Πολλές φορές μια στρατηγική πολιτικού χαρακτήρα μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ανθρωπιστική παρέμβαση, μια προσπάθεια αυτού του είδους. Και είχαμε και το παράδειγμα του εκπροσώπου της Ούρα που είπε ότι εκεί που δεν έχει γίνει πραγματικά πρόοδος είναι το πολιτικό ε, θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε περισσότερο για το σημείο αυτό. Δεν θα μας κάνετε μια πρόταση η οποία αν θυμηθούμε τη διπλωματική ιστορία της Υπήρου μας μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μας οδηγεί σε νέες σκέψεις. λέτε πέρα από την ανάγκη περιεκτικότητας που τονίζεται, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε περισσότερο με τον αραβικό σύνδεσμο. Μια λύση λοιπόν <clears throat> που θέλει να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται ήδη αυτή η κίνηση, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει με τον αραβικό σύνδεσμο και όχι μόνο. Αλλά φυσικά θα παίξει σημαντικό ρόλο το Συμβούλιο των Χωρών του Πεσκού Κόλπου, και ο αραβικό Σύνδεσμος ιδιαίτερο ρόλο. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα επίση Και τρίτον, ήσασταν κάπως επιφυλακτικός για δύο θέματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα φώτα της επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο. <clears throat> Πρώτο ερώτημα είναι το ερώτημα που αφορά το καθεστώ του Μπασάρ Αλασάντ. Λέτε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε ο αγώνας κατά του Ισλαμικού κράτους δεν θα ενισχύσει τον Μπασαρά Ε, συναντήσαμε τον κύριο Μιτσουά σήμερα. Δεν μιστούρα, ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει πραγματικά ένα τέτοιο κίνδυνο. Θα μπορούσατε να μα πείτε κάτι περισσότερο, γιατί ιδίω λέτε ότι ο πραγματικό κίνδυνο είναι η αντιπαράθεση Σουνιτών και Σιητών. Και τέλο, αν πάμε προ την κατεύθυνση αυτή, και αναπτυχθεί μια πολιτική αυτού του είδους, θα πρέπει να μας πείτε και ποια είναι η άποψή σας και για το Ιράν, που η θέση τους παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην περιοχή. Μιλήσατε για τους Χεσμολά, αλλά η στάση του Ιράν θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, πρώτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παγκόσμια στρατηγική. Αυτό είναι ουσιαστικό να φτάσουμε στο τέλος να είμαστε συνεπεί. Δεύτερον, τι θα κάνουμε να δούμε με ποιον θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όπως είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος και το τρίτο είναι το θέμα του Μπασάρα Λασάντ και του ρόλου του Ιράν που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ κύριε Πεγιώνο, κύριος Ντόνζον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας καθηγητά και εγώ προσπογράφω απόλυτα αυτά που είπε ο Βανσάν Πεγιόν. Θα ήθελα όμω να εστιάσω περισσότερο το θέμα της πολιτικής εξόδου από τις περιοχές αυτές τις τόσο βασανισμένες της Συρίας και του Ιράκ. Έχετε μιλήσει για μια περιεκτική λύση, μια πολιτική λύση η οποία θα είναι περιεκτική και στη Λιβύη. Αυτή είναι η μαγική λέξη, είναι η λέξη που είναι λιγάκι του σειρμού. Δεν το λέω αυτό αρνητικά. Το ερώτημά μου εδώ είναι κατά πόσον οι ομάδες αυτές θέλουν να βρούνε μια περιεκτική λύση, μια πολιτική ε, περιεκτική λύση ή τουλάχιστον λιγότερο σεχταριστική λύση, όπως στην περίπτωση του Ιράκ, θα μπορέσει να μειώσει την στρατολόγηση από το Ισλαμικό κράτος. Τα τελευταία χρόνια, με μια λιγότερο σεχταριστική πολιτική του Ιράκ, δεν υπήρξε μια τέτοια δεν θα είχε υπάρξει αν είχε υπήρχε μια τέτοια πολιτική η ανάδυση και πάλι του Ισλαμικού κράτους που υπήρχε ήδη από την εποχή του Αζαρκαουή αν δεν υπήρχαν λοιπόν όλοι αυτοί οι τομείς, τα στρώματα και οι φυλές που θεωρούσαν ότι είναι αποκλεισμένοι από την λειτουργία του κράτους. Αλλά ο σκληρός πυρήνας αυτής ομάδας που έχει μια καλή σημαντική παρουσία στις χώρες αυτές το ερώτημα είναι θέλει μια πολιτική λύση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιδεολογικό του καλούπι παραμένει η μονοπόληση της εξουσίας και όχι ο διαμερασμός της εξουσίας και εάν δεν ασκήσουν το μονοπόλιο της εξουσίας σε αυτά τα εδάφη θα προτιμούσαν να έχουν ένα μικρό κομμάτι όλου αυτού του εδάφους της επικράτειας όπου de facto ασκούν πλήρως την εξουσία τους. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι πραγματικά εφικτή μια περιεκτική λύση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε τρομοκρατικέ ομάδε. Ευχαριστώ. Κύριο Παντσέρη. Μα πιέζει ο χρόνο, οπότε και εγώ θέλω να σα πω το εξή μόνο. Να μην πούμε για τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, ε, είναι γνωστά. Αλλά αυτά τα οποία μας ε, τόνισε ο εισηγητής. Ε, εκεί θέλω να σταθώ. Μήπως τώρα Κάνω μια τρύπα στον που μιλάμε για, για την παρέμβασή μας, για αυτές τις χώρες εκεί που συνεχίζεται η, αναμέτρηση και συνεχίζεται και η αναρχία σε αυτές τις χώρες που η οποία οδηγεί όταν υπάρχουν και αυτές οι διάφορες ομάδες. Άρα, μας τα είπατε πάρα πολύ ρεαλιστικά, πώς έχει το τοπίο. Και θα πρέπει να προσέξουμε την επιχειρηματολογία για αυτές τις χώρες. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε καμία συνέπεια στην πολιτική της αυτά τα χρόνια. Να. Έτσι έδειξε τι προβλήματα έχουμε. Και κάτι άλλο ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε μία ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουμε σε επιμέρους χώρες με τις διμερείς τους σχέσεις. Και ε, το κίνητρό τους είναι περισσότερο η, η, η, παρά κάτι άλλο, παρά τα δικαιώματα. Επομένως, ξαναγυρίζουμε στο ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική που σήμερα δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο τώρα, πολύ σύντομα. Δεν ξέρω τι πρεσβεύεται. Αλλά εδώ έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε το οποίο είναι έτσι ψυχολογικού χαρακτήρα. Το πώς θα ερμηνευτεί αυτού του είδους η, κουλτούρα που διαδίδεται με, το Ισλαμικό κράτος. Το, ότι τελικά αυτοί προβάλλουν ό,τι φοβίζει περισσότερο. Την μητέρα όλων των φόβων, το φόβο του θανάτου. Και από την άλλη μεριά σε αυτό το επίπεδο εμείς βρισκόμαστε σε αδύναμη θέση. Είπαμε για ζώνη απαγόρευση πτήσεων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κύριε καθηγητά Βαρπέλη για τη συστάση σας. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο στην πρώτη παράγραφο και στην έκτη. Στην πρώτη παράγραφο γράφεται ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την πολιτική τάξη αφενός και τα ανθρώπινα δικαιώματα αφετέρου. Και ότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος, ενδεχομένως να υπήρχε, στην Ευρώπη να απαιτούμε προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, που υπονομεύουν την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, πράγμα που θα έχει ως ε, επίπτωση το χάος και την κατάρρευση. Στην παράγραφο 6 λέτε να συνεργαστούν περισσότερο οι μυστικές υπηρεσίες και με τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου, της Λιβύης, των κράτων του Περσικού κόλπου ναι, βεβαίω θα πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίε και να συλλέγουμε, αλλά πού είναι τα benchmark, τα ορόσημα. Τουλάχιστον το περασμένο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Υπουργών Εξωτερικών είπε ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει με κάθε τίμημα και είστε και επιστήμον. Ε, και αν θέλετε περιστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποια είναι αυτά. Δεν το λέω με κινησμό, γιατί θα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τι θα κάνουμε, να επιτρέπονται τα βασανιστήρια, ολίγα βασανιστήρια, ε, ή ε, χρησιμοποιούν ε, πληροφορίες ε, που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες αποσπάσει μετά από βασανιστήρια. Και αυτά τα δικά μας κράτη δικαίου τα ε, ευλογούν μετά την 11η Σεπτεμβρίου είδαμε ότι είχαμε περισσότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν οδήγησαν σε περισσότερη ασφάλεια, μάλλον το αντίθετο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λοχπίλερ. Η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που μας παρέχει πολύ χρήσιμες και πάρα πολύ εύστοχες αναλύσεις εκτίμησα πάρα πολύ τα διάφορα στοιχεία που εξειδικεύσατε, τη χρηματοδότηση, τη στρατολόγηση των νέων. Θα ήθελα όμως να επιμείνω στο εξή. Τώρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αρχίζω από το μακροπρόθεσμο. Σημειώνω ότι μέσω μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει την ορθή προσέγγιση. Να υποστηρίξουμε την οικοδόμηση κρατών δικαίου, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σταθεροποίηση της Μεσογείου. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει κατευθυντήρια γραμμή μας. Από την άλλη όμως βράχει πρόθεσμα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πιο αποτελεσματική και πιο αποφασιστική δράση. Σημειώνω αυτό που είπατε, να συνεργαστούμε περισσότερο με τον Αραβικό Σύνδεσμο ιδιαίτερα έτσι ώστε να αναπτύξει εκείνο ίδιο μηχανισμό ειρήνης και ασφάλειας. Πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση. Πριν όμως θα πρέπει να υπάρχει και εντολή από πλευρά των αραβικών κρατών αλλά και βούληση να εργαστούν επ' αυτών. Είχε ήρθει εδώ στις 19 Ιανουαρίου Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Ναμπίλ Αλάραμπι, και επανειλημμένα τόνισε ότι ε, σκοπός και αποστολή του Αραβικού Συνδέσμου είναι να συνεργάζονται ε, για πολιτιστικά και θρησκευτικά θέματα και όχι πολιτικά. Πώς θα δοθεί όθηση λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Και δεύτερον, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ε, ριζοσπαστικοποίησης αυτής της ενώ Χρειάζονται πιο χειροπιαστές ε, προσπάθειες και συγκεκριμένες και σας ερωτώ πώς μπορούμε καλύτερα να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές. Κάποιες από τις χώρες Μέση Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν ε, ε, ενδιαφέροντα προγράμματα το Μαρόκο ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη θεολογική εκπαίδευση των ημάμιδων. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε όμως σε ποιο επίπεδο για να εξασφαλίσουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Και ποιο ρόλο εκεί βλέπετε ε, για την Ευρωμεσογειακή Ένωση που προς το παρόν θα μπορούσε να ξαναγίνει ένα θεσμός που θα παίζει ρόλο κλειδί. Έχω και άλλες δύο ερωτήσεις. Το τρίτο στοιχείο αφορά τη Λιβύη. Σημειώνω αυτό που αναφέρεται για τη μόνιμη ομάδα επαφής που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αραβικές χώρες για να υποστηρίζεται η δράση της Ένωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα και πολύ σημαντική. Έτσι ώστε η Λιβύη να μην γίνει μια δεύτερη Συρία εκεί. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν το αναφέρατε καθόλου. Πώς βλέπετε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αραβικού Συνδέσμου και Αφρικανικής Ένωσης. Διότι ας μην λησμονούμε ότι υπάρχει Σαχέλ και κίνδυνος διάδοσης και επιμόλυνσης στην υπόλοιπη Αφρικανική Ήπειρο. Θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάμις. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να ακούσω την απάντηση που θα δώσετε στον κύριο Πελιών για την ε, θέση του Ασάτ στη Συρία και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Μιστούρα. Από ό,τι βλέπω δεν πηγαίνουν πολύ, δεν πάει πολύ μακριά. Και ποιές είναι και εναλλακτικέ λύσεις γιατί πάρα πολλά εξαρτώνται από αυτό το οποίο θα συμβεί στη Συρία. Και πάλι είναι ένας χώρος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απούσα. Οικονομικά ήταν παρούσα αλλά δεν είχε καμία απόλυτη επιρροή. Και στο Λίβανο το ίδιο πράγμα. Αναφερθήκατε στο σημαντικό παράγοντα των Εσβολά που κατά κάποιο τρόπο συγκρατεί το Ισλαμικό κράτος. <clears throat> Πώς βλέπετε όμως να είναι οι δυνατότητες για μια προσέγγιση με το Ιράκ. Και δεδομένου ότι η Εσβολά αρχίζει να γίνεται ρεχοκοκαλιά του Λιβανικού στρατού και ένα σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση του Λιβανικού έθνους. Πώς θα επηρεάσει αυτό. Και επίσης, μήπως μπορούμε ως Ευρώπη να συνεχίσουμε να παραγνωρίσουμε την ε, αντιπαράθεση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Εμείς τώρα που ήμασταν στο Λίβανο και στην Ιορδανία μας είπαν όλοι αν εξακολουθείτε να παραγνωρίζετε αυτή τη σύγκρουση δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει την ε, Αλνούσα ως ένα παρακλάδι ένα παρακλάδι κατά κάποιο τρόπο του Ισλαμικού κράτους του Ντάς. Και θεωρεί ότι είναι και αυτό ένα, ένα δημιούργημα, μια επινόηση της δύση. Και τέλος η Λιβύη. Η Λιβύη είναι μια σαφής περίπτωση όπου η Ευρώπη ήταν απούσα και δεν έχει δράσει. Μετά από τη στρατιωτική επιχείρηση που επέτυχε τους στόχους της, και τους στόχους του λιβικού λαού και αυτό δεν θέλω να το παραγνωρίσω. Ήταν μια περίπτωση όπου η Ευρώπη δεν λειτουργήσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Κοινοβούλιο μας ζήτησε από την αρχή μια αποστολή της ε, ΚΕΠΑ να τονίσει την ε, ευρωπαϊκή διάσταση και αυτό δεν έγινε. Και τώρα μας λέτε ότι έχουμε όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη, δημιουργία ε, έθνους, συμφιλίωση κτλ. Τίποτα από αυτά δεν χρησιμοποίησαμε. Και δεν νομίζω ότι και πάλι είμαστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουμε. Απλώ υπάρχει ανταγωνισμό των κρατών μελών λόγω οικονομικών συμφερόντων. Ξέροντα ότι αυτό μα έφερε εδώ που είμαστε. Είναι πολύ φανερό ότι αυτή η κατάσταση τη κατάρρευση των κρατικών δομών και του να είναι καταφύγιο η Λιβύη για τους τρομοκράτες, αυτό θα μπορούσε να το προβλέψει κανείς από πολύ παλιότερα αν πρόκειται να λειτουργήσουμε και με άλλους συνομιλητές και ο Αραβικός Σύνδεσμος μπορεί να είναι ένα σημαντικός εταίρος, αλλά έχει και τα ωριά του ο Αραβικός Σύνδεσμος, όπως είπαν οι Είμαστε όμως σαφείς σε σχέση με το ποιον το κοινό μας συμφέρον θα δουλέψουμε ως Ευρωπαίοι ή όχι. Αν δω τι γίνεται στο Ιράκ, είναι αποτρόπαιος ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη-μέλη μας. Αυτοί που είχαν παίξει ρόλο στρατιωτικό δεν θέλουν να συντονιστούν μεταξύ τους. Οι καημένοι πεσπεργάδες δεν έχουν καν το στρατιωτικό εξοπλισμό. Βλέπετε ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν κανένα απόλυτο, απόλυτα ρόλο. Δεν λειτουργεί τίποτα στους καταβλισμούς <clears throat> του Ιράκ ε, ή, της, ε, ή του Λιβάνου που έχουμε 300.000 παιδιά τα οποία δεν πήγαν στο σχολείο. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα έφορο έδαφος για, την, ε, για τον προσυλλητισμό τρομοκρατών. Δεν γίνεται μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΚΟ, της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Κομισιόν, καμία μορφή συντονισμού. Τίποτα δεν γίνεται για μακροχρόνια αρρωγή για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι έχουν ένα μέλλον. Και αυτό αφορά ιδίω τους κατοίκους του Ιράκ. Πού βρισκόμαστε λοιπόν και τι θα κρατημέλει. Ευχαριστώ Άννα. Κύριε Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που είπε η κυρία Γκόμες θα μπορούσα να τα πω και εγώ. Σα ευχαριστώ κύριε καθηγητά για τη μελέτη που μας παρουσιάσατε και δεν θέλω να σα επικρίνω με αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σύγχυση αυτή η μελέτη, όπως έχει μεγάλη σύγχυση και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αυτή μια επικίνδυνη φράση. Θα πρέπει εδώ να είμαστε πιο σαφείς τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ομάδα κρατών μελών και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Το είδαμε σε όλη αυτή την περιοχή ότι διαφορετικά κράτη-μέλη ασχολούνται με διαφορετικό τρόπο και ακολουθούν διαφορετικά σενάρια. Αλλά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι για το τι μπορούμε να πετύχουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτό σημαίνει ουσιαστικά μία ε, εγγυημένη αδράνεια. Γιατί θα πετάει ο ένα τον παλάκι στον άλλο. <clears throat> Τρία συγκεκριμένα σημεία. Για το σημείο 4 που είπατε, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συλλογική της δράση θα πρέπει να συντονίζεται με τη δράση του Αραβικού Συνδέσμου. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, αμφιβάλλω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική μια τέτοια αντιμετώπιση. Κανείς στον αραβικό κόσμο δεν θεωρεί τον Αραβικό Σύνδεσμο ένα σημαντικό πολιτικό οργανισμό πέραν του διαλόγου. Στο σημείο 7 επίσης κάντε μια έκκληση να σταματήσει η τσιγαθιστική προπαγάνδα στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε μαζικά την ελευθερία του λόγου και θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη νομοθεσία που μας εξασφαλίζει αυτά που θέλουμε κυρίως, αλλά κύρια μου, αντίρρηση είναι για το σημείο 3 για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν κανονισμού για τη λειτουργία και τη δράση όλων των θρησκευτικών οργανισμών και αντίστοιχων μη κυβερνητικών οργανισμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να φύγει αμέσω αυτό από το κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια πιο εμπριστική δήλωση, μια δήλωση η οποία θα οδηγήσει σε μεγάλη αντιπαράθεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν περιορίσουμε για μια μονάχα ομολογία την θρησκευτική ελευθερία, αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα σε όλη τη μουσουλμανική κοινότητα. Κατανοώ ότι αυτό είναι ένα προσχέδιο. Σα ευχαριστώ για τι ενδιαφέρουσε προτάσει αλλά για το σημείο 3 θέλω να σα ζητήσω αμέσω να αφαιρεθεί από το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Σμιθ. ο κύριο Χριστέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά και κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Το Ισλαμικό κράτος έχει υποστεί απώλειες μετά τις επιδρομές και ε, τις επιθέσεις της συμμαχίας. Αλλά στρατολογεί και νέους τώρα ε, περισσότερους και ανακυκλώνει τους ανθρωπίνους πόρους, ακόμα και την ηγεσία του. Και ε, ασκεί και πολιτική. Γνωρίζουμε ότι μια ιδεολογία δεν την πολεμάς με στρατό απέναντι με τα όπλα. Σήμερα συζητούμε τρόπους πολιτικής επίλυσης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε ακριβώς τις ακραίες εξεμιστικές ιδεολογίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Και πώς θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας εκεί στην περιοχή. Εσείς ε, προτείνατε συγκεκριμένα μέτρα, ιδιαίτερα πολιτικά, αλλά υπάρχουν και άλλα, οικονομικά ενδεχομένως, που θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα όφιλε να υιοθετήσει. Έχω μια ερώτηση που θα ήθελα να ε, συνδέσω με την επόμενη συζήτηση που θα έχουμε για την αναθεώρηση πολιτικής γειτονίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Θα πρέπει να είναι πιο ισχυρό το πλαίσιο ασφαλείας και ε, να αποτελέσει ενδεχομένως μια σπίδα ή μια λύση ε, των κρατών της Ένωσης αλλά και της γειτονίας. Ευχαριστώ κύριος Καστάλτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει στα Ισπανικά κύριος Καστάλτο. Συγχαρητήρια κύριε Δόκτρα Βαρέλη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγησή σας και, να σας ακούσουμε. Και θα ήθελα τώρα κάτι να, να πω όσον αφορά τις σκέψεις μας εκθέσατε ε, για να μπούμε λίγο σε βάθος μας. Είπατε πρώτα πρώτα για τις πηγές, ε, τις χρηματικές, τις οικονομικές που έχουν οι Ισλαμιστές και είπαμε ότι τώρα έχουν ασχοληθεί και επικοινωνούν δεν, δεν, δεν μεταφράζεται στην άντληση του πετρελαίου. Όμως είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φήμες που κυκλοφορούν και σε σχέση με το τι γίνεται, ότι τουλάχιστον, τουλάχιστον λένε ότι υπάρχει ανοχή, τουλάχιστον ανοχή από πλευρά των κρατών του κόλπου. Και από την άλλη μεριά λέμε και για χρήματα τα οποία λαμβάνουν αυτοί. Ε, και τα χρήματα τα οποία πήρανε στην αρχή του εμφυλίου πόλεμου στην Συρία. Τώρα τι γίνεται για να αποφύγουν το, το ότι κάποιοι μπορούν, θα θα πάνε και θα στείλουν χρήματα από τον Περσικό κόλφο. Έχουμε τρόπους να τους σταματήσουμε. Ή μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή ευρωπαικη να λάβει κάποια πιο αποφασιστικά μέτρα. Και αυτό ισχύει και για τη χρηματοδότηση από πλευρά τη Τουρκία. Μα είπατε για τη σχέση Αλγάιντα και Ισλαμικό κράτο. Μα είπατε στην αρχή για ε, συνύπαρξη ανταγωνιστική. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά ε, ακριβέ. Από την άλλη μεριά όμω συνεχίζει να ισχύει το ότι έχει αποδείξει το Ισλαμικό κράτος ότι είναι πολύ πιο ε, αποτελεσματικό. Είδατε τι έγινε ε, ότι προσπάθησαν ε, να στήσουν ένα κράτος με αυτό το μοντέλο του Χαλιφάτου και ήταν πολύ πιο ελκυστική για τον κόσμο. Εκεί που στο έδαφος που ελέγχουν σε Συρία και Ιράκ και πόσο προσπαθούν να χτίσουν ένα κράτος αυταρχικό, βίο, αλλά είδαμε ότι έκαναν ένα ούτως πιν ποιοτικό άλμα σε σχέση με αυτό που έκανε η Αλκάιδα. Άρα το ερώτημα είναι το εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε την υποστήριξη των διαφόρων φυλών στο Ισλαμικό κράτος. Γιατί αυτό ήταν πολύ βασικό όσον αφορά την ενίσχυση του Χαλιφάτου και την επέκταση του ελέγχου που έχουν πάνω στο, ε, στην περιοχή εκείνη. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από αυτό που κάνουμε τώρα. Επίσης, σχέσεις με τις άλλες ε, τρομοκρατικές οργανώσεις στην Λιβύη. Μας είπατε κάποια εθνικά στοιχεία, είπατε ότι ίσως είναι 2.000, ίσως είναι 3.000, ε, αλλά έχουμε και την ε, ε Αλσαρία που είπαμε ότι φτάνει το 10.000 Ακριβώς όπως είπατε και με το οποίο συμφωνώ, να δούμε εμείς πώς θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε, και, αλλά να αποφύγουμε αυτό να τους ενώσει, αντί να είναι διερημένοι μεταξύ τους. Άρα πρώτα πρώτα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις πρώτες δύο φατρίες, τον Μπρουκ και από την άλλη μεριά την Τρίπολη. Γιατί δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μόνο τη μία πλευρά, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε αποτυχία. Γιατί εδώ πέρα μιλούμε για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που δεν εκπροσωπούνται από εκείνη την ε, πλευρά. Και να, πώς βρίσκουν οι Ισλαμιστές το έφορο έδαφος για στρατολόγηση. Γιατί δεν μπορούμε να ασχέσουμε την ε, προπαγάνδα με άλλη προπαγάνδα αλλά μπορούμε να τη σταματήσουμε με ένα πολιτικό σχέδιο, πολιτικό πρόγραμμα σοβαρό. Ανάληψη πολιτικής δράσης που να έχει συνοχή με κάποιες ε, στέρες, συνεπείς ε, θέσεις, μελετημένες ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονομένα τα κρατη Αλλά επίσης έτσι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει η ριζοσπαστικοποίηση και αυτά να, να το προχωρήσουμε χέρι-χέρι και παραλλήλως. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Το πρόβλημα είναι ο κύριο Βαρβέλη. Θα χρειαστεί δύο ώρες τώρα για να σα απαντήσει όλα αυτά που τον ρωτάτε. Κύριο Σπανιό, παρακαλώ. Ε, πρόεδρε, σύντομα, γιατί περνάει και η ώρα. Θα ήθελα να ε, πω πόσο εύστοχα τα είπατε και θα χαιρετίζω αυτό κύριε καθηγητά. Ε, η Λιβύη ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη ε, ως ανάχωμα και είναι ξεχωριστή η θέση της ως προς τον ΤΑΕΣ και ως βάση στα μετόπιστεν. Παρά τα διάφορα ερωτήματα και τα αιτήματα και ορισμένοι ζητούν στρατιωτική επέμβαση εκεί, θα ήθελα να θυμίσω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσο αφορά όλα αυτά. Εσείς μιλάτε για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με μία μόνιμη επιτροπή, ένα θεσμικό όργανο ανάμεσα στους Λιβύους και τους τοπικούς ε, παράγοντες που είναι ε, Αλγερία, Κατάρ, ε, Μαρόκο, Τινσία, Αίγυπτος, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι μια εναλλακτική λύση, μια προοπτική που θα πρέπει να βρούμε εμείς και να εκτάσουμε ως ευρωβουλευτές απέναντι σε διάφορους υπερβολικά θερμοκέφαλου και πολεμοχαρείς κατά την άποψή μου. Και σε σχέση με όλα αυτά και την ευρύτερη περιοχή, ε, θα ήθελα να πω ότι πολλοί πιστεύουμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ε, συνοδευτικός. Το είπε και ο Πεγιό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους τοπικούς αραβικούς φορείς. Ε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα αραβικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μάρτιο του 2013 αυτό το αποφάσισε ο Αραβικό Σύνδεσμος. Δύο χρόνια έχουν περάσει. Το Μάρτιο του 2013 και ακόμα περιμένουμε να δημιουργηθεί αυτό το δικαστήριο και έχει προταθεί να εδρεύει και στο Μπαχρέιν μάλιστα. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας σχετικά. Και μια τελευταία πρόταση, παρατήρηση ε, συμφωνώ απολύτως με την μελέτη σας εκεί που λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει την μουσουλμανική κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές. Το είπε και η κυρία Γκαμπριέλ. Είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, να διευκολύνουμε το διαθρησκευτικό διάλογο και να ε, ε, εκπαιδεύσουμε και ε, κληρικούς μουσουλμάνους στη χώρα μας. Ο Μπερνάρ Κασνεύ, υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, προτείνει να διπλασιαστούν οι θέσεις εκπαίδευση στα πανεπιστήμια της ε, Γαλλίας σε θεολογικές σχολές μουσουλμανικές. Ε, ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας. Ευχαριστώ κύριε Πεγιόν. Ο κύριος Χάν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ομιλητή μας. κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση επιδεινώνεται. Έτσι δεν είναι σε σχέση με σε αυτές τις ομάδες. Είχαμε πρώτα τους Ταλιμπάν, μετά την Αλκάιντα και τώρα τον Ταές. Συνεχώς οξύνεται και φαίνεται ο, κάθε καινούριος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Και δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο στο κείμενό σας έχετε αντιμετωπίσει τη ρίζα του κακού. Πού οφείλονται όλα αυτά, για ποιο λόγο ε, έχουμε αυτή την κλιμάκωση της βίας και κάθε κύκλος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Ε, ποια είναι λοιπόν τα λάθη. Ε, πολλές από τις κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν στους λαούς τους τη συμμετοχή στα κοινά. Και αυτό είναι ένα θέμα και είναι ε, μία από τις αιτίε που οδηγεί σε αυτές τις ακραίες ομάδες που εμφανίζονται. Αναφερθήκατε κάπως ακροθυγώς στο Ιράν. Η επιρροή του Ιράν ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο εμείς ε, αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε. Δεν είναι μόνο το Ιράκ, ο Λίβανος και η Σύρια. Και πάλι τι συμπέρασμα έχετε εξαγάγει και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε να διευκολύνουμε τις σχέσεις Ιράν με Σαουδική Αραβία ε, για να βρούμε και τα μερίσματα ειρήνης που αναζητούμε εκεί. Και ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε και για το δικό μας ρόλο στις χώρες αυτές. Το ανέφεραν πολύ οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Μήπως είναι πολύ πιο εύκολο να πας εκεί και να ρίξεις ένα δικτάτορα. Αλλά η ανοικοδόμηση ε, ενός ε, χρεοκοπημένου, κατεστραμμένου κράτους είναι πολύ πιο μακροχρόνια και πολύ πιο επίπονη και δεν βοηθάει, δεν αρκεί λοιπόν η κατάρριψη ενός καθεστώτος. Και ένα τελευταίο έχει να κάνει με όλο αυτό το αφήγημα. Έχει μεγάλη σημασία να μην επιτρέψουμε ε, στις χώρες εκεί της περιοχής να ε, συγχαίουν τα πράγματα. Ε, γιατί κάπως ε, χρησιμοποιούν όλη αυτή την ιστορία για να σκληρύνουν την καταστολή τους. Και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες στην περιοχή που μπορεί να είναι μεν Ισλαμιστές, αλλά είναι ειρηνικοί ε, και δεν ε, ευαγγελίζονται τη βία, αλλά μια απάντηση στον Ντάες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Τελευταίος, ο κύριος Κόρβιν Μίκε, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Είναι σωστό όταν σας λέω ότι αν δεν είχε ανατραπεί ο Σαντάμ Χουσέιν και δεν είχε υποσκαφθεί η εξουσία του Μασάρα σαν δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στην περιοχή. Ο κύριος Μπαρδέλη έχει το λόγο. Παρακαλώ σύντομα. Σας ευχαριστώ για όλε αυτέ τι ερωτήσει σα για να απαντήσω σε όλου. Ε, θα, θα, θα, θα, πάρα πολύ ώρα αλλά πρώτα πρώτα θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι ε, δυσεπίλητα, υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα, δεν επιλύονται αυτά, δεν επιλύονται ούτε για μια συγκεκριμένη χώρα, ε, ας πούμε για μια, από μια Ιταλία, μια Γαλλία, μια Γερμανία, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Επομένως εμείς οι πανεπιστημιακοί οφείλουμε να κάνουμε απλώς αυτό το policy prescription και να ξέρουμε πού είναι τα όρια των δυσκολιών και οπότε σας εκθέτουν πως είναι τα ζητήματα και ξέρουν πόσο δύσκολο να λυθούν οι αποφάσεις και ξέρουν τις περισσότερες φορές ότι το, το, το timing της διπλωματίας δεν είναι το timing το οποίο έχει ένας πολιτικός για να λάβει κάποιες αποφάσεις για να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει κοινή γνώμη. Αν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την κοινή γνώμη σε τόσες χώρες που είναι σε κατάσταση έξελη σε σχέση με την επέκταση του, του, του, του Ισλαμισμού, της μετανάστευσης ε, αυτό το ζήτημα του ριζοσπαστισμού, ε, για το τι γίνεται με τις ε, ντόπιε σε κάθε κράτος Ισλαμικές κοινότητες. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ευφυείς απαντήσεις ό,τι γίνεται, όπου γίνεται αυτό. Οπότε θα πρέπει να σας τονίσω ότι βασικό θέμα το οποίο τώρα χαρακτηρίζει αυτό το πολύπλοκο τοπίο στη Μέση Ανατολή είναι, είναι το ίδιο το τοπίο της, ε, το, το, δηλαδή ότι χρειάζεται να έχουμε κάποια σύνθεση θέσεων ε, των πιο σημαντικών από τους ε, εμπλεκόμενους. Οπότε και εμείς ως Δύση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να πούμε στους άλλους εσείς σταματήστε να φαγώνεστε ενώ ούτε εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κοινέ θέσεις. Και αυτό σας το λέω διότι αφορά και το Ιράκ αλλά αφορά και την Λιβύη. Η Λιβύη ένα τέτοιο παράδειγμα. Μας δείχνει το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Γιατί κάθε ε, κράτος, παράγοντας της τοπικής διεθνούς σκηνής, ε, πάει σε κάποιο μια τέτοιο διαπραγμάτευση, μια τέτοιο μετασχηματισμό. Και αυτό γίνεται από το κομμάτι του κράτους το οποίο έχει την πλειοψηφία και, ε, και έχει τέλο αυτό το, το plan B. Ε, και είναι αυτό το οποίο ακριβώς τώρα συμβαίνει στην Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και στα Εμμυράτα που υποστηρίζουν το τον Μπρουκ και τον ε, στρατηγό Αφτάρ. Το δε Κατάρε, Τουρκία και άλλες χώρες που υπεστήριξαν την κυβέρνηση της ε, Τρυπόλεως. Οπότε δεν συμφωνούμε. Απλώς ευνοούμε τη μία πλευρά εις βάθος της άλλης. Και βέβαια είναι και το θέμα τώρα της νομιμότητας. Ε, άλλοτε το λαμβάνει υπόψη, άλλοτε όχι. Στην Λιβύη πολύ λιγότερο. Γιατί είχαμε αυτές όλες τις εκλογές στην ε, Λιβύη και είδαμε πως οι μετέσχοντες και πιο δύσκολη και είδαμε ότι τελικά είχαμε αυτή την κυβέρνηση, είχαμε και τι έγινε μετά με, με, με, με αυτούς που ανέλαβαν τα ενία της χώρας από το Τομπρούκ που τελικά δεν έχουν την νομιμότητα της πλειοψηφίας του λαού. Και πάντα λέμε στις μελέτες για το nation building, state building, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι μπορούμε έτσι να βρούμε τη λύση για την Λιβύη. Οι Λίβοι να δώσουν τη λύση για τη χώρα τους, αλλά αυτό είναι λίγο υποκριτικό, γιατί είδατε τι έγινε ε, από τα χρόνια του, από τα χρόνια του Καντάφη τι προέκυψε στη συνέχεια. Κάναμε από τότε λάθος. Όμως δεν είναι Ευρωπαίοι οι Λίβοι. Άρα θα πρέπει πρώτα που να βρουν την ε, ταυτότητά τους θα πρέπει να βρουν ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο και να μην ε, πόλεμα ένα στον άλλο. Αυτό το οποίο έγινε εκεί δεν ήταν μια ε, επανάσταση. Ήταν ε, ένας ξεσηκωμός μια φατρίας έναντι της άλλης. Επρόκειτο για εμφύλιο πόλεμο. Θα πρέπει να το ε, αναγνωρίσουμε, να τους βοηθήσουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Οπότε θα πρέπει πρώτα να τεθεί ένα τέρμα εκεί και να ξεκινήσει ένα συγκρότηση του κράτους ή του έθνους, state building που λέμε κλπ. Αλλά όχι να γίνουν πρώτα οι εκλογές και να μην έχει προηγηθεί ένα συγκρότηση του κράτους, η οικοδόμηση του έθνους. Είδαμε τι έγινε το 2000-2003 και με το Ιράκ. Πριν δοθεί κάποια επίφαση νομιμότητα σε κάποια κυβέρνηση, είδαμε ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα έπρεπε να, έχουν, να τα έχουν βρει και να έχουν πετύχει τη σταθεροποίηση της χώρας τους. Αυτά γενικώ τώρα για να δούμε για κάποιες επικρίσεις που διατυπώθηκαν. Όχι, κανείς δεν είναι κατά της θετικής ελευθερίας φυσικά και αυτό είναι βασικό και για μένα και για τους συναδέλφους. Εάν κάτι τέτοιο φάνηκε, όχι το διαψεύδουμε. Οπότε αυτό το οποίο θέλουμε εδώ είναι να καταγράψουμε το πώς οι Ισλαμικές ευρωπαϊκές κοινότητες θα πρέπει να εμπλακούν για στη διαχείριση του προβλήματος της ευρωπαϊκής ασφάλειας σε κάθε επιμέρους χώρα. Ε, γιατί πρώτα-πρώτα είναι προς το δικό τους συμφέρον. Το δικό τους συμφέρον δεν είναι να προβάλλονται και να φαίνονται ως τρομοκράτες και να τους κατηγορούν ότι είναι τρομοκράτες. Άρα χρειάζεται συνεργασία με το κράτος. Αυτό όμως δεν πάει να πει άρση της θρησκευτικής ελευθερίας. Βεβαίω και δεν μιλούμε τώρα για χρήση βασανιστήριων. Είπαμε για συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών. Εγώ δεν είμαι ειδικό και δεν μπορώ να πω ακριβώ πώ θα γίνει αυτή η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε χρήση βία, χρήση βασανιστήριων. Είπαμε όμως ότι θα πρέπει τώρα να μπουν κάποιες νέες προτεραιότητες όσον αφορά την ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πολλές φορές παραμένει χωρίς μεγάλη ισορροπία όσον αφορά από τη μια μεριά την εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και δεν, δεν υπάρχει κάποιο ουσιώδες περιεχόμενο σε αυτά τα οποία εξαγγέλει η, η Ένωση. Για άλλα το πειρατήσατε, είπατε για το διεθνές κοινικό Βεβαίω είπαμε ότι μπορεί στο να, στην ε, διαμόρφωση της διεθνούς κοινής να λάβουμε υπόψη το Ιράν. Είναι πολύ ισχυρός παράγον και αν θέλουμε η ειρήνη στην Μέση Ανατολή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρουσία ενός παράγοντα τόσο σημαντικού όπως το Ιράν. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ στο Ιράν και αλλάζουν συνεχώς την τελευταία περίοδο. Οπότε είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλέξει και το Ιράν μέσω της διεθνούς κοινότητας. Να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο. Πέραν του να υποστηρίζουμε την κάθε επιμέρους ε, απόφαση που λαμβάνει το Ιράν. Αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Όπως έγινε για τις πιο σημαντικές κρίσεις Όπω ε, όπως έγινε για το Ιράκ, όπως έγινε για τη Συρία, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, είναι πολύ σημαντικός παράγον και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Ο, τώρα μιλήσατε για τη συμπερίληψη, για τις πολιτικές της συμπερίληψης, όσον αφορά και τις δυνατότητες συμφωνίας. Ε, όχι βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι στο τραπέζι να βραντεύουν να κάτσουν και οι τζιχαντιστές. Αυτοί είναι σαφώς τρομοκράτες. Ε, τίποτα τέτοιο δεν μπορεί να εννοούμε. Αλλά μιλούμε για συμπερίληψη κάποιων κοινοτήτων που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υποστηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Δηλαδή κάτι το οποίο ε, σταματάει το χάος το οποίο υπάρχει, το οποίο οδήγησε στην άνοδο των Ισλαμιστών. Είδατε, ε, είπαμε ότι έχουμε αυτά τα, τα χρεοκοπημένα κράτη, τα κράτη που χρεοκοπούν. Ε, όπου έχουμε τέτοια κράτη, τότε έχουμε την άνοδο της ε, τρομοκρατίας και του τζιχαντισμού. Η Εμένη, Νιγηρία, ε, Σαχέλ, Λιβύη, Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν. Ε, αυτό πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο να το σχεδιάσει κανείς, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να το υλοποιήσει. Αλλά πάντως νομίζω ότι χωρίς μια τέτοια πολιτική ε, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι. Και κυρίως μακρόπνο. Δεν μπορούν να αποσπάσουν τίποτα αποτελέσματα για τη Λιβύη τώρα. Δεν νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορούσαμε να λάβουμε μια αυθεντική πρωτοβουλία μεσολάβησης ε, διαμέσου των επιμέρους μελών. Ε, πρωτοβουλία δηλαδή, Λεόν, πρωτοβουλία ΟΗΕ. Με πολλοί είναι οι κίνδυνοι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει εδώ πέρα ο κίνδυνος ε, της ανάφλεξης. Γι' αυτό και θα είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτή τη συμφωνία μεταξύ των μερών peacekeeping, διατήρηση της ε, ειρήνης. Αυτό θα πρέπει να είναι ο άμεσος στόχος. Γιατί από την άλλη μεριά έχουμε τους παραστρατιωτικούς, έχουμε τους διάφορους ένοπλους, τις διάφορες ομάδες. Οπότε είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Αλλά τουλάχιστον να ανακάτουν γύρω από το τραπέζι οι πιο, ε, πιο σημαντικές ομάδες ακόμα και να έχουμε συγκεκριμένες ε, κυρώσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα αυτό θα μπορούσε να γίνει από την διεθνή κοινότητα. Γιατί υπάρχουν εκεί κάποια, κάποια κόμματα, κάποιες παρατάξεις που δεν θέλουν να ειρηνεύσει η χώρα. Αυτοί θα μπορούσαν να υποστούν κάποιες κυρώσεις. Να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέτρα δυνατόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για να δούμε πώς Α, η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος πρώτα-πρώτα σκητάει το εθνικό της συμφέρον. Καλά το κάνει. Σωστή δίκιο έχει. Αλλά έχει κάπως διαφορετική οπτική των πραγμάτων από αυτή που έχουμε εμείς. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οπωσδήποτε η υποστήριξη της Άφταρ, η υποστήριξη του, του, του, των Ισλαμιστών, αυτό έχουν κάνει και αυτό είναι επικίνδυνο οπότε αν έτσι τους υποστηρίξουν τότε θα καταλήξουν όπως έγινε και στη Λιβύη σε ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο θα κατησχίσει και είδαμε τι έγινε και τελικά κατέληξε σε επανάσταση και ξεσηκωμό που είχαμε στην Αραβική Άνοιξη και έτσι έχουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και άρα δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα και θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση όλης της Μέσης Ανατολής και οδήγησαν σε όλον αυτόν τον φονταμεταλισμό και στο χαλιφάτο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαρδέλη για την εμβάθυνσή σας στο τόσο σημαντικό και πολύπλοκο αυτό θέμα. Θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν λάβει το λόγο και ευχόμαστε καλή πτυχία στον κύριο Πεγιού και αφήνω στον κύριο Πλένκοβιτ στην Προεδρία για το επόμενο σημείο. Dear colleagues, let's... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ερχόμαστε στο πέμπτο σημείο της μέσης διάταξης, δημόσια ακρόαση για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Είναι το πρώτο βήμα <clears throat> προς την κατεύθυνση της ε, έκθεσης που θα παρουσιάσει ο Έντουαρτ Κούκαν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην ακρόαση που έγινε ε, του Επιτρόπου Χάν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Χάν ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν του ζήτησε να κάνει μια αναθεώρηση της πολιτικής, μια επισκόπηση και αναθεώρηση της πολιτικής μέσα στον πρώτο χρόνο της εντολής της Νέας Κομισιόν. Στις 4 Μαρτίου η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα παρουσιάσουν ένα πράσινο έγγραφο σε σχέση με τη διαδικασία αυτή αναθεώρηση η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική δράση μετά θα κάνουν διαβουλεύσει με όλου του εμπλεκόμενου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, θα, και τα άλλα όργανα και θα παρουσιάσουν ένα τελικό έγγραφο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει να συμβάλλει με τις δικές του διαβουλεύσεις και την έκθεση πρωτοβουλία του κ. Κούκαν. Η πολιτική γειτονία ξεκίνησε το 2004 από την Επιτροπή Πρόν με το στόχο να μην υπάρξουν άλλε διαχωριστικέ γραμμέ μεταξύ τη διευρυμένη Ευρώπη και των γειτόνων τη. Ο στόχο ήταν να υπάρξει ένα τόξο τόξος και ένας δακτύλιος φύλων με <clears throat> κοινέ βάσει, αλλά όχι κατά ανάγκη κοινού θεσμού. Έτσι έχει εμπλουτιστεί μια πολιτική η οποία ήταν καταρχήν διμερής με μια πολύ ε, μερή διάσταση όπως η πολιτική της ε, Βαρκελόνης, και η, η Ένωση για τη Μεσόγειο, η Στατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα και η Πολιτική για την Ανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερα έχει τονιστεί πρόσφατα η ανεπάρκεια αυτής της πολιτικής και των εργαλείων τους. Ήταν ιδιαίτερα άκαμπτη για να αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις και παρά το υψηλό επίπεδο οικονομικής υποστήριξης έδειξαν τα γεγονότα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τη δημιουργία πιο σταθερών δημοκρατικών κοινωνιών η Αραβική Άνοιξη το 2011 και τα επακόλουθά της οδήγησαν σε μια αναθεώρηση αυτής της πολιτικής με μεγαλύτερη <clears throat> εστίαση στην πρόθεση βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας που να συμπεριλαμβάνει περιεκτική οικονομική ανάπτυξη. Έλαβε επίση αυτή η αναθεώρηση το γεγονό ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσει για να ισχύσει η αρχή του περισσότερα για περισσότερα. Και ζητά επίσης την συμπερίληψη και τη κοινωνία των πολιτών. Μετά από την αναθεώρηση όμως του 2012 υπάρχουν νέες εξελίξεις και στα νότια και στα ανατολικά της Ευρώπης, όχι μόνο η κρίση στην Συρία, Λιβύη και την Ουκρανία, αλλά και η αυξανόμενη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, άλλων παικτών που παρέχουν εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν η στιγμή της επισκόψης είναι επίκαιρη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει ποιε είναι οι αξίες επί τη βάση των οποίων εργάζεται και να καθορίσει τις προτεραιότητες στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων τους. Θα πρέπει να διαφοροποιήσει τους εταίρους σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα, τα επίπεδα ανάπτυξής τους, τις προτεραιότητες αυτών των ιδίων και να προτείνει ένα επίπεδο διαλόγου που να αντιστοιχεί σε όλα αυτά χωρίς να υποσκάψει τις αξίες επί των οποίων βασίζεται η ενέργειά μα. Σήμερα έχουμε δύο εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα παρουσιάσουν τι μελέτε που έχουν συντάξει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κρίνουν την πολιτική γειτονία και θα παρουσιάσουν και προτάσει για το μέλλον. Έχω την ε, χαρά να παρουσιάσω τον κύριο Γρηγόριο Γκρομάτσκι από το Ινστιτούτο <clears throat> Δημοσίων Υποθέσεων τη Πολωνία, ο οποίο έχει συγγράψει τη μελέτη ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση μετά από πέντε χρόνια και Ρώσια Αναθέωση και τον κύριο Χάσα Μαζάν από το, από Πανεπιστήμιο του Κάιρο στην Αίγυπτο που θα παρουσιάσει τη μελέτη του για την ε, αξιολόγηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της νότιας γειτονίας της. Είδα και την ομιλία του Επιτρόπου Χάν στην Βιέννη, τα τέσσερα σημεία που παρουσίασε, διαφοροποίηση, συμμετοχή, εστίαση και ευκαμψία και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ναι. Ε, σας παρακαλώ να παραμείνουμε στα 10 λεπτά γιατί κάπως έχουμε καθυστερήσει με τα προηγούμενα θέματα συζήτησης ιδίως το τελευταίο το οποίο ήταν ιδιαίτερα συν, συνδεόμενο με το ζήτημα αυτό και μετά από την παρουσίασή σας θα είναι ο Έντουαρ Κούκαν ο οποίος θα λάβει πρώτο το λόγο και μετά οι άλλοι σκιώδει εισηγητέ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Γκρομάσκι. Thank you, <coughs> Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την ανατολική εταιρική σχέση και θα σας παρακαλούσα να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα εξή τρία πράγματα. Ε, την περασμένη πεταετία ε, της πολιτικής αυτής ε, την προοπτική κατά δεύτερο λόγο μετά από δύο-τρία χρόνια και τέλος ε, δυνατότητες πολιτικής, επιλογές και συστάσεις. Ε, Το πρώτο, εξιολόγηση της περίοδου μέχρι τώρα. Ξέρουμε ποια είναι η διαφορετικότητα, υπάρχει και ο ρωσικός παράγοντας και τέλος ε, να σας πω κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις. Πρώτον, κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ήταν ο ελάχιστο κοινό παρονομαστή που θα μπορούσαν να δεχθούν όλα τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης το 2009. Η μια πολιτική μας προς Ανατολάς. Η ε, ε, ανατολική γειτονία είναι ένα στοιχείο που διακρίνει την πολιτική γειτονία και την αντιπαραβάλλει προς την νότια. Η ανατολική γειτονία ε, ήταν ένα αποτελεσματικό πακέτο, μια δέσμη πάρα πολύ αποτελεσματικών ε, προτάσεων και μέτρων. Ε, υπεγράφει η Συμφωνία Σύνδεσης με την DCFTA το 2006 δημιουργήθηκε προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια και τέλος, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, άρχισε υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων για να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτε των χωρών αυτών. Ε, στην Ουκρανία και τη Μολδαβία επίσης είχαν προταθεί εν μέρη κάποια στοιχεία από αυτά πριν την Ανατολική Γειτονία. Ε, έχουν μεγάλες διαφορές οι έξι χώρες. Το είδαμε αυτό το 2009 όταν ξεκίνησε η πολιτική αυτή και παραμένουν σαφέστατες για να μην πω μεγαλύτερες ακόμα στις αρχές του 2015. Δύο υποομάδες μπορούμε εκεί να διακρίνουμε, υποσύνολα. Πρώτον, ε, χώρες με αυταρχικές κυβερνήσεις και δεύτερον χώρες που είναι δημοκρατικές σε ένα σημαντικό βαθμό. Η πρώτη ομάδα κρατών περιλαμβάνει Αζερβαϊτζάν και Λευκορωσία και η δεύτερη Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία. Η Αρμενία είναι κάπου στη μέση, πιο κοντά ε, προς τη δεύτερη όμως, την πιο δημοκρατική ομάδα. Ο ρωσικός παράγων τώρα επανειλημμένα ακούγεται ότι η Ρωσία είναι κατά της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Όχι μόνο αυτό, είναι και κατά της Συμφωνίας Σύνδεσης των χωρών της γειτονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία θεωρεί ότι είναι κενό γράμμα αυτό το θέμα της γειτονίας γιατί δεν πρόκειται ποτέ χωρίς να μπουν στην Ένωση. Αυτό φάνηκε το 2013 στις διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία ε, και ε, την Αρμενία. Και άλλαξε δραματικά τότε η ε, στάση της Ρωσίας. Έρχομαι τώρα στα επιτεύγματα και τις ελλείψεις και αδυναμίες. Τρία είναι τα πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα, συμφωνίες σύνδεσης, και ε, ελευθέρων συναλλαγών, ε, άρση θεωρήση διαβατηρίων με τη ε, Μολδαβία και ενεργειακή ένωση με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Παρ' όλα αυτά, περιορίζεται σε τρεις μόνο χώρες και όχι στο σύνολο των έξι κρατών που αποτελούν την Ανατολική γειτονία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ε, καλύτερα από ό,τι ελπίζαμε και παρά τις πιέσεις της Ρωσίας ε, έχουν καμφθεί οι αρχικές αμφιβολίες και από πλευράς της Ένωσης και από πλευράς των χωρών αυτών για τις διμερείς σχέσεις. Οι διμερείς σχέσεις μας είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από μία πενταετία. Οι διμερείς σχέσεις μπορούν κατά την άποψή μου να θεωρηθούν ως μερική επιτυχία για τρεις χώρες, ενώ η πολυμερής διάσταση θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον ε, ως ε, αδυναμία ή οπισθοχώρηση. Ε, ποια είναι τώρα η προοπτική για την επόμενη διετία-τριετία. Ο ρωσικό παράγων στο μέλλον, η θέση Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρε που έχουν καλύτερε επιδόσει, που είναι η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία, και οι επιδόσει των υπολείπων. Πάμε πρώτα στη Ρωσία. η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί να εμποδίζει ε, την ε, προσέγγιση στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα η πολιτική του Πούτιν ε, και λόγω της οικονομικής κρίσης θα συνεχίσει να παραβιάζει και να τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των χώρων αυτών την επόμενη χρονιά. Το πιο πιθανό είναι η Ουκρανία να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από τη Ρωσία ως ειδική περίπτωση και να εξακολουθήσει η Μόσχα να ε, αποσταθεροποιεί την Ουκρανία για να μην υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση του Κιέβου με την Ουκρανία ποντάρει αυτό για να ε, υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στη σημερινή κυβέρνηση. Ποια είναι η θέση τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει σφήνα ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. E αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική μας πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Ε, Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι τα πραγματικά συμφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της και των μεμονωμένων κρατών μελών απέναντι στη Ρωσία. Στο εσωτερικό της Ένωσης υπάρχουν ε, διάφορες σκέψεις από την ε, ε, detente, την εξομάλυνση και τευνασμό με κάθε τίμημα μέχρι τα πιο επιθετικά σχόλια θα πρέπει, όχι μόνο στην Ουκρανία μας ενδιαφέρει να επικρατήσει η δημοκρατία, αλλά σε όλες τις χώρες. Οι εντάσεις μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας θα πρέπει να ειδωθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ε, που είναι ε, ε, αυτή η διελκυστίδα ανάμεσα στην φιλελεύθερη δημοκρατία και το σύγχρονο αυταρκισμό οι χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις χρειάζεται ακόμα να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι ελίτ και οι πολιτικές και οι οικονομικές στις τρεις χώρες που ανέφερα, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, ε, παραμένουν μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ακόμα και αν υπάρχουν ευρωπαϊκές, φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που είναι σημαντικές, υπάρχουν και άλλοι όμως που του συμφέρει περισσότερο το status quo. Therefore, Γι' αυτό η κοινωνία θα παραμείνει παράγον κλειδί για τις μεταρρυθμίσεις στη Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία. Μόνο ε, αν δεν χαλαρώσει η πίεση από το λαό που θα ε, απαιτεί εκδημοκρατισμό και τη ε, δημιουργία ενός κράτους που θα λειτουργεί βάσει των κανόνων του κράτους δικαίου, θα θέσουν τα θεμέλια για τις ε, μεταρρυθμίσει. Έρχομαι τώρα στο Αζερβαϊτζάν και στη Λευκορωσία. Οι πρόεδροι Αλίεφ και Λουκασέκο δεν πρόκειται να δεχθούν δημοκρατικέ μεταρρυθμίσεις. Αυτοί θέλουν να διατηρήσουν εκεί την αυταρχική τους ε, εξουσία. Έχουν αλλάξει και οι δύο τα συντάγματα των χωρών τους για να είναι διαβίου πρόεδροι. Are Έχουν στήσει πολιτικά συστήματα που δεν ε, συνάδουν με την δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία. Και το τελευταίο, ε, συστάσεις και ε, που είναι ανοιχτά για τη πολιτική μετά από τις νέες ε, πραγματικότητες και επαναξιολόγηση ή επανεξέταση της ε, πολιτικής ανατολικής γειτονίας. Ένας ανοιχτός γεωπολιτικός ανταγωνισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας έχει αρχίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, περιμένει κρίση στη σχέση της με τη Ρωσία που θα διαρκήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εποχής του Πούτιν. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε μια έξυπνη στρατηγική αποτροπής της συγκράτησης της Ρωσίας. Οι κυρώσεις παραμένουν ο κορμός της πολιτικής απέναντι στην Ένωση και είναι ε, μια κύρωση για περιορισμό των ζημιών και όχι πανάκια για αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων με τη Ρωσία πρόθεσμα και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις μέχρι ότου η... δεν πρέπει να αρθούν μέχρι ότου επανέλθει η Κρυμαία στην Ουκρανία και η Ρωσία σταματήσει την επεκτατική της δράση. Η ρωσική ελίτ Ε, λαμβάνει υπόψη μόνο τη συνέπεια στην πολιτική. Αν δει το ρωσικό καθεστώς ότι υπάρχει επιταλάντευση, αυτό θα ορθεί ως δείγμα ανδυναμίας. Πέραν της επίθεσης Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει αλλάξει εκ βάθρων την κατάσταση το 2014 που είναι μια διάκριση μεταξύ τριών χωρών που έχουν ήδη υπογράψει μια συμφωνία στα πλαίσια του DCFTA και πλησιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και η Λευκορωσία δεν θα υπογράψουν συμφωνία σύνδεσης μέσα στα πλαίσια του, του DCFTA στο ορατό μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπονήσει μια στρατηγική για να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. και οι εταιρικέ αυτές σχέσεις μέσα στην πολιτική γειτονία. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων πέντε ετών, είναι σαφές ότι η αρχική σύλληψη του 2009 δεν είναι πλέον πλησίων της πραγματικότητας της αρχής του 2015. Χρειάζονται σημαντικές τροποποίησεις. Μια αναθεωρημένη πολιτική γειτονία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη πολιτική ε, πτυχή και όχι ένα τεχνικό εγχείρημα όπως είναι σήμερα. Η σταθεροποίηση της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι ο πιο σημαντικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον. Το να διαχωρίσουμε τις χώρες της γειτονίας σε δύο ομάδες είναι απαραίτητο. Οι... Αυτές που υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης και αυτές Λευκορωσία, Αζερβαϊτζάν και Αρμένια. Αρμενία που δεν το έχουν κάνει. αρχή περισσότερα, για περισσότερο θα πρέπει να τηρηθεί. Αλλά η συνορική αντιμετώπιση της πολιτικής γειτονίας που περιλαμβάνει και την ε, φιλελευθεροποίηση στις προξενικές θεωρήσεις και όχι μόνο την εταιρική σχέση σε οικονομικά θέματα πρέπει να μείνει ανοιχτή για όλες και τις έξι χώρες. Για την Πελαρούς, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην κοινωνία των χωρών αυτών και όχι να κάνουμε μη ρεαλιστικές ε, προτάσεις συνεργασία με το Μίνσκ, το Γερεβάν και το Μπακού. Η συνεδρίαση κορυφής της, ε, Ευρω... της ε, πολιτικής γειτονίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένας σημαντικός διάβλος συνεργασίας, αλλά θα πρέπει να είναι σε δύο κομμάτια πρώτον με τις χώρες που έχουν κάνει συμφωνία σύνδεσης και το δεύτερο τμήμα και με τις έξι χώρες. Οι διμερείς σχέσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο για την κοινωνία και των έξι χωρών. Εν τέλει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, διτό τέτοιο ρόλο υποστηρίζοντας τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας για να συμπεριλάβουν το κοινοτικό κεκτημένο στο νομικό σύστημα των χωρών τους. Ε, αυτό θα είναι ένα βήμα το οποίο θα έχει σημαντική ε, σημασία για την εφαρμογή της πλήρους συμφωνίας ελευθερού εμπορίου και τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μεταλαμβαδεύσουν την εμπειρία του στα κοινοβούλια αυτών των τριών χωρών σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και, την, και των ομάδων πιέσεων. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκραμάτσκι. Παραμείνετε σχεδόν στα 12,5 λεπτά. Σας ευχαριστούμε για τις ε, προτάσεις. Ο κύριος Μαζέν έχει το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή μας η μελέτη προετοιμάστηκε από τον υποφαινόμενο τον που Μπουμαζέ και θα σας πω για τέσσερα σήμερα πρώτα πρώτα. Πόσο αποτελεσματική είναι τα χρηματοδοτικά, χρηματοοικονομικά μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμπληρωματικότητα επίση τη πολιτική τη Ένωση με την πολιτική των κρατών μελών για την πολιτική γειτονία προ Νότον. Αλλά επίση και πώ όλα αυτά διαπλέγονται με το τι κάνουν οι υπόλοιποι παράγοντε, για να δούμε τι συστάσεις διατυπώθηκαν κατόπιν της ε, ε, μελέτης. Για να δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής σήμερα. Αυτής της πολιτικής. Έχουμε δει τα αρνητικά, αλλά υπάρχουν και κάποια θετικές περιοχές στην πολιτική σας. Θα πρέπει αυτά να λυθουν υποψη υπόψη πρώτα-πρώτα ό,τι προκύπτει από τα έγγραφα και από κάποιες διαδικασίες. Και επίσης, τι ισχύει όσον αφορά την ε, κυριαρχική ευθύνη. Και όλα αυτά σε σχέση με τα όσα είχαμε ως μέσα πολιτική προηγουμένως αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι στερούνται κριτικής αυτές οι πολιτικές πρώτα-πρώτα. Τα προβλήματα που είχε η πολιτική προς Ανατολάς. γιατί πρώτα πρώτα σχεδιάστηκε για την γειτνία της Ανατολάς και κατόπιν για την γειτνία της Νότον, που είναι διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετική ιστορία. Οπότε και οι κοινοτικές πολιτικές για την γετνίαση τελικά οδηγούσαν προς Ανατολάς στην προσχώρηση κάποιων χωρών, αλλά αυτό δεν ισχύει για την προς Νότο γετνίαση. Και αν κάποιες χώρες θέλουν να είναι μέλη κάποιες περιφερειακές οργάνωσεις, αυτή η οργάνωση δεν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για να δούμε τα έγγραφα από τον οποίο προκύπτει πώς σχεδιάστηκε αυτή η πολιτική κοινωνία, Ε, υπερβολικά φιλόδοξη καταρχήν και οι επιμέρους φιλοδοξίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Επίσης τα θέματα ευημερίας, σταθερότητας, ασφάλειας βλέπουμε ότι είναι περίπλοκες οι διαδικασίες μετασχηματισμού στον Νότο και βλέπουμε επίσης ότι πολλές φορές άλλο μεταρρύθμιση και άλλο σταθεροποίηση και πολλές φορές όλα παίρνει εις βάρος της ευημερίας. Άρα χρειάζεται να τεθούν κάποιες προτεραιότητες και μια που έχω τις ρίζες μου σε εκείνη την περιοχή δεν μπορούμε τους στόχους όλους να τους επιδιώξουμε ταυτόχρονα. Επίσης, το να μην υπάρχει αμοιβαία απόδοση ευθύνη. Αυτό είναι παραπλανητικό. Γιατί τους καλούμε να είναι υπόλογοι των πραξιών τους. Αλλά εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο προς εμάς. Θετικό αυτό ως έννοια, αλλά δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Τώρα, η στήριξη της δημοκρατίας. Στην πολιτική επιστήμη γνωρίζουμε ότι στις ε, φτωχές χώρες είναι σύντομη ζωή της δημοκρατίας, οπότε θα μας εκπλήξει για το ότι εκεί προς και στις πρώτες αυτές χώρες ε, έχουμε φτώχεια και ένας τρόπος να υποστήριξουμε την δημοκρατία είναι να τους βοηθήσουμε οικονομικά. Να στηρίξουμε τις οικονομίες τους. Ξέρω ότι και αυτά είναι συζητήσιμα, αλλά πολλοί πολιτικοί επιστήμονες θα συμφωνούσαν και θα λέγανε μερικοί από αυτούς ότι υπάρχει κάποιο είδους κατόφλι ε, για κατακεφαλήν εισόδημα πάνω από το οποίο μπορεί να πιάσει, να ριζώσει η δημοκρατία. κάνει κάποια βήματα η δημοκρατία, αλλά είναι τόσο πιο δύσκολη η κατάσταση όσο πιο φτωχή είναι μια τέτοια χώρα. Άρα να, αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Τώρα επίσης όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό είναι το ότι θεωρείται ότι τα πράγματα κυρίως εξαρτούνται από την προσφορά και όχι από τη συζήτηση. Το 2011 είδαμε ότι τότε υπήρχε ζήτηση για δημοκρατία. Προέρχομαι από εκεί και σας ε, διαβεβαιώ ότι τα πράγματα είναι έτσι. Τώρα, σήμερα, σήμερα ακούσατε τι είπε ο εισηγητής για το Ισλαμικό κράτος. Έχουμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα σταθερότητας και ασφάλειας. Σταθερότητα πάντως έχει υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική θεματολογία. Γι' αυτό και λέμε για αναθεώρηση της πολιτικής γετινίασης. Γιατί άλλα πράγματα ίσχυαν το 2011 που σχεδιάστηκε η πολιτική, προς νότον δηλαδή. Να, για παράδειγμα, να σας πω με στοιχεία. Έχουμε ένα γκάλο που το χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε σε όλες, σχεδόν όλες τις χώρες ε, της πολιτικής γυμνίασης και ρωτήσαμε τι είναι το ιδανικό, τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε οικονομική βοήθεια, είπαν όλοι. Δεν, δεν θέλουν καμιά πολιτική στήριξη και παρέμβαση. Θέλανε η μεταρρύθμιση έτσι να γίνει προς οικονομικής και να, γίνει βαθμία και όχι απότομα με ριζοσπαστικό τρόπο. Να ρίξετε μια ματιά. Γιατί έτσι μπορείτε να δείτε μια εικόνα του τοπίου. Το πώς βλέπει ο κόσμος η ιδιωδός τα πράγματα. Πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε κατά τον κόσμο. Τώρα τι γίνεται με τα άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρία μη. υπήρξε μια περιορισμένη πρόοδος. Υπήρξαν εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας με το Μαρόκο, την Τινησία και την Ιορδανία, αλλά όταν πρόκειται για τα χρήματα, τα χρήματα τα οποία είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υλοποιήθηκαν, ήταν περιορισμένα. Δεν βοήθησε και η αστάθεια της περιοχής αλλά είναι γεγονός ότι σε επίπεδο χρηματικής υποστήριξης η πρόοδος ήταν πολύ περιορισμένη. Αν συγκρίνει κανείς και το μερίδιο κατά κεφαλήν των χρημάτων που δίνεται στο νότιο τμήμα της Μεσογείου εναντί της ανατολικής πλευράς της ε, Ευρώπης, πέραν των Παλαιστινιακών εδαφών, βλέπει κανείς ότι η υποστήριξη προς τον νότο είναι πολύ μικρότερη. 5,2 ευρώ κατά κεφαλή ενώ είναι 6,9 στο ανατολικό τμήμα της, στα ανατολικά της Ευρώπης, η διαδικασία τώρα επισκόπησης και αναθεώρησης. Θα πρέπει να συμμετέχουν και περισσότεροι. Γίνεται μια αρχική διατύπωση, μετά η κάθε χώρα καλείται να σχολιάσει, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι στην αρχή και δεν θα πρέπει να υπεραπλοποιήσουμε την διαδικασία μετάβασης η οποία είναι πολύπλοκη, έχει τα πάνω της και τα κάτω της και δεν μπορούμε να την αξιολογούμε μονάχα με ένα κατάλογο ε, σημείων που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη μορφή των μεταβάσεων. Και υπάρχει και περιορισμένη ικανότητα αντικτύπου και σε οικονομικό επίπεδο Μπορεί να σας φαίνονται πολλά τα χρήματα αυτά, αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν να δώσουν οικονομική βοήθεια, αυτά είναι μικρά ποσά, ιδίως σε σχέση με τη βοήθεια του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Εκεί είναι μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Έρχονται πιο γρήγορα τα χρήματα, δεν υπάρχει ερεσιμότητα τόσο έντονη σε πολιτικό επίπεδο και επομένως επηρεάζουν περισσότερο. περιορισμένου όντου του χρόνου, θα προχωρήσω παραπάνω σύντομα σε ό,τι αφορά τα θέματα τη συμπληρωματικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών. Ανεφέρθη προηγουμένω από κάποιου έντιμου βουλευτέ ότι υπάρχουν ανισομέρειε και αντιφάσει πολλέ φορέ περισσότερο σε ό,τι αφορά τι χώρε του Νότου, ακόμα και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις, όχι και μεταξύ μονάχα των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορές μηνυμάτων σε ό,τι αφορά σχετικά τις διαφορετικές θέσεις για τη Λιβύη, αυτές που αναφέρθηκαν από τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου και αυτές από τον, την υπατή εκπρόσωπο. Ο στόχος ήταν η προστασία των ε, αμάχων. Υπήρξε και έλλειψη συντονισμού μεταξύ Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερη από ό,τι έπρεπε χρηματοδότηση της εταιρική σχέση για τη δημοκρατία. Και τώρα αν συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους ξένους παίκτες, και εδώ εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θεωρούν όλοι ότι είναι τμήμα της Δύσης, ότι είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι κρίμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι σε, οικονομικούς, σε πολιτικούς όρους, αλλά σε οικονομικούς όρους και άλλους όρους αντιμετωπίζεται θετικά στον αραβικό κόσμο. Θεωρείται ως η Ήπειρος η οποία μπόρεσε να ξεπεράσει τις εσωτερικές της διαφορές είναι ένα υπόδειγμα περιφερειακής ολοκλήρωσης που όλοι στον αραβικό κόσμο θα ήθελαν να ακολουθήσουν με, με θόνο. Αλλά η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπλέει πάντα με, την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι μόνο εκ των υστέρων και μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε σε ό,τι αφορά πολλές από τις κρίσεις στην Αραβική Άνοιξη και ακολούθησε κατά πόδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραγματικά η περίπτωση Αιγύπτου είναι ένα παράδειγμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά παραμένουν η πιο ισχυρή δύναμη σε επίπεδο ασφαλείας στην περιοχή και σε μια περιοχή που η ασφάλεια είναι η μεγαλύτερη μέρημνα, ο ρόλος των Πολιτείων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε και για τα κράτη του Περσικού κόλπου. <clears throat> Έχει τη μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη και δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα να σταθεροποιηθούν οι χώρε τη Μεσογείου χωρί το Συμβουλίο Συνεργασία του Περσικού Κόλπου. Λυπάμαι τώρα, τώρα δεν προφταίνω. Συστάσει, μόνο δύο διαφάνειε έχω. Πρέπει να κατανοήσουμε το ότι η ασφάλεια γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα. Η ασφάλεια και όχι μεταρρυθμίσει είναι η πρώτη προτεραιότητα τη περιοχή και πρέπει να το κατανοήσουν οι βουλευτέ. Χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερο προπολογισμό για το 2014-2020 αλλά με πιο στοχευμένο τρόπο. Οι εταίροι από την νότια οχτή της Μεσογείου πρέπει να πάρουν τι σωστέ ε, αποφάσει και ζητούν εμπειρογνώμονε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνουν επενδύσει στον πολιτισμικό διάλογο και του ελέγχου στα σύνορα να υποστηριχθούν τα καταβλισμοί προσφύγων στην Ιορδανία και το Λίβανο. Πρέπει να εργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους εταίρους. Δεν είναι μοναχα η γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η γειτονιά άλλων περιφερειακών δυνάμεων όπως το Συμβούλιο συνεργασία του Περσικού Κόλπου. Πρέπει να σταθεροποιηθεί η περιοχή και να ενισχυθούν οι οικονομίες τους και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συνεκτικότητας των απόψεων και των δηλώσεων να μην υπάρχουν πολλαπλά μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Dr. Ευχαριστώ πάρα πολύ καθηγητά. Θα δώσω μέσα στο λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Εντουαρτ Κούκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν μπω στην ουσία, ένα τεχνικό θέμα που έχω να πω. Έχω το πρόγραμμα της ακρόασης εδώ που σημειώνει ότι αρχίζει στις 5 και άρχισε η ακρόαση 45 λεπτά αργότερα. Ε, Αντρέη, εγώ σε εκτιμώ ως πρόεδρο, αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης. Ε, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης των αξιότιμων προσκεκλημών μας. Ε, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι δίκαιο. Το λέω για να αποφευθεί στο μέλλον τέτοια κατάσταση. Αν έρχεται κάποιος να προεδρεύσει εκτός ΑΦΕΤ, θα πρέπει να ενημερώνει η γραμματεία τον εκάστοτε την εκάστοτε πρόεδρο ότι υπάρχουν και κανόνες. Ακόμα, εντάξει, αν είναι 5-10 λεπτά πάει στο καλό, αλλά 45 λεπτά, 3 τέταρτα δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος που μας απασχολεί. Πρώτον, Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για τη συνεισφορά τους ε, για την αναθεώρηση ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αυτό που μου άρεσε στις παρουσιάσεις σας ήταν ότι και οι δύο αναλύσεις που κάνατε δεν είναι ακαδημαϊκές, θεωρητικές, αλλά πραγματικά ασχολούνται με το ζήτημα. Είναι ουσιαστικές και ε, περιλαμβάνουν και πολλές ε, καλές ιδέες και πολλά ε, καλά μηνύματα. The report. Και θα πρέπει να ε, τις ε, συμπεριλάβουμε στις εργασίες μας για την εκπόνηση της έκθεσης για την αναθεώρηση. Νομίζω ότι ήταν πολύ τα όσα μας είπατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, χαίρομαι που σου ζητούμε τα ευρωπαϊκά θεσματικά όργανα, την πολιτική γειτονία. Θα πρέπει να τη διορθώσουμε. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ε, προβλήματα και προκλήσεις που έχουμε ε, στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η Επιτροπή μας ε, ασχολείται και έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια ξανά και ξανά με τις εξελίξεις της χώρας γειτονίας και προσβλέπω και στη δική σας συνεργασία, στη συνεχή αναθεώρηση, να μας βοηθήσει να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο. Ε, από τις παρουσιάσεις που ακούσαμε σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι σαφές ότι πρόκειται για διαφορετικές εξελίξεις. Αλλά συχνά τα προβλήματα είναι παρόμοια. Οι περισσότερες χώρες της γειτονίας, για διάφορους λόγους, είναι σε μια κρίσιμη καμπή ή για να το πω αλλιώ, είναι αρκετά εύθραυστη η κατάσταση, ε, ευμετάβλητη, σε βαθμό που διαφέρει από χώρα σε χώρα και επικύλει. Χρειάζεται για τη σταθεροποίηση, οικονομική ανάπτυξη και δημοκρατική εξέλιξη και εμείς έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό στην πολιτική γειτονία. Επειδή και όσο διαφορετικά και ε, να είναι τα αίτια των προβλημάτων, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά εργαλεία για να βοηθήσουμε τους τέρους μας έτσι ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι. Οι εξελίξεις τελευταίας πενταετίας μας έκαναν να αναθεωρούμε την πολιτική γειτονία. Λαμβάνοντας υπόψη και άλλους εξωγενείς παράγοντες και αντιμετωπίζοντας νέες πραγματικότητες. Στην ανατολική γειτονία είμαστε αντιμέτωποι με νέες πραγματικότητες και νέες προκλήσεις. Το ε, είπε ο καθηγητής Ζοντάσκη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και οφείλεται στην πολιτική της Ρωσίας στην περιοχή. Όλο και περισσότερο καθίσταται σαφές ότι ε, πρόκειται για διαφορετικές ε, χώρες, κάθε φορά διαφορετικές ομάδες, που έχουν και κειμενό με διαφορετική προθυμία συνεργασίας και ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε πολύ ωραία. Στον Νότο, μετά την ε, Αραβική Άνοιξη, προβληματιστήκαμε τι θα κάνουμε και τι κάνει κανείς με μια αναπτυσσόμενη χώρα που είναι σε μεταβατική εποχή. Και πάλι οι διαδικασίες ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους και πολύ συχνά αποκλίνουν από τον αρχικό στόχο. Οι συστάσεις για πιο ευέλικτη και διαφοροποιημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών θα είναι σημαντική για μας στόχη κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης. Ωστόσο δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε τις αρχές που εντάξαμε πριν από κάποια χρόνια στην πολιτική γειτονία. Όπως περισσότερα για περισσότερα ή λιγότερα για λιγότερα. Η προθυμία λοιπόν των κρατών να μπουν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις απαιτητικές θα πρέπει να υποστηρίζεται αντιστοίχως και να ανταμείβεται. Μακροπρόθεσμα είμαστε προσιλωμένοι στην πολιτική γειτονία και δεσμευμένοι. Ε, ωστόσο, η πολιτική θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά στις ταχείες εξελίξεις και αλλαγές που Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα εργαλεία πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας για την πολιτική γειτονίας και να προετοιμαστούμε για να χρησιμοποιούμε πιο σωστά, πιο αρμόζοντα και πιο ταχεία καμιά φορά μέσα, ε, κατά περίπτωση, ε, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις οι συμβιβασμού στι βασικές αρχές και αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι και κόκκινη γραμμή αυτή, με όλη την ευελιξία και ό,τι άλλο θέλετε. Συμπέρασμα. Σε ό,τι αφορά τη δική μου έκθεση, θα ήθελα να δούμε και ποια είναι η πολιτική μας, το πλαίσιο, αλλά και ποια είναι τα μέσα και τα εργαλεία. Θα κοιτάξω τις προτεραιότητές μας και την εκτίμηση ε, και τι άποψη έχουν οι χώρες της και του Νότου. Αυτό ήθελα να μιλήσω, να πω Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω γενικά, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, για κάθε πτυχή, για κάθε θέμα της πολιτικής γειτονίας, διότι δεν του παρόντος. Έχουμε καιρό, αν δείτε το χρονοδιάγραμμα μέχρι να εγκριθεί η έκθεση, θα γίνουν πολλές συζητήσει ακόμα ε, για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, Ομιλητέ μα, θα μα προβληματίσουν αυτά που μα είπατε και θα τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Είστε Κριστέα. κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε για την εισαγωγή που κάνετε στο θέμα αλλά και για τους δύο μιλητές. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της έκθεσης ε, Κούκαν από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών. Και πολύ θετικό ότι σήμερα κάναμε την ακρόαση. Έχοντα υπόψη επομένω τα δύο έγγραφα και ακούγοντα και εσά, βλέπουμε ποιε είναι οι δύο απειλέ και για την Ανατολή και για τον Νότο. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να αναθεωρήσουμε την πολιτική γειτονία σε πλευρά ε, στόχων, μέσων, εμπλεκομένων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τις ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αναφερθήκατε όλοι στο θέμα της ε, ε, ε, ασφάλειας γιατί ακριβώς τώρα έχουμε όλες αυτές τις συγκρούσεις προ και προς και προς Νότον. Οπότε βεβαίως έχουμε κάποιε κάποιες φιλοδοξίες αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τα θέματα ασφάλειας, να μην τα αποσυνδέουμε γιατί κάναμε κάποιες παράλληλες κινήσεις αλλά ακόμα και εκτός της ε, εντολής της ε, πολιτικής γειτονίασης θα πρέπει να έχουμε ε, ένα κράτος που να λειτουργεί εύρυθμα δεν υπάρχουν και κάποιες αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και σας ρωτώ, πώς θεωρείτε ότι η ε, ασφάλεια μπορεί να καλυφθεί καλύτερα από μια αναθεωρημένη πολιτική κοινωνίαση, γιατί με διαφορετικούς τρόπους και οι δύο μας ε, αναφέρατε τη λογική της διεύνησης στην ε, πολιτική κοινωνίαση και κάνατε τη διάκριση μεταξύ πολιτικής και τεχνικής αντιμετώπισης. Κάνετε κάποιο διαχωρισμό ανάλογα με φιλοδοξία και επιδόσεις και επίσης μας είπατε ότι θέλετε συγκεκριμένου τομείς ε, να δείτε τα πράγματα ε, από οικονομική σκοπιά. Άρα τι θα γίνει, μια προσέγγιση από το Α μέχρι το Ω επί τη βάση της εμπειρίας, της διεύρυνσης και έτσι να προχωρήσουμε για όλη την ε, πολιτική γειτονίαση συνολικά, κράτος δικαίου, σύγχρονοι θεσμοί, όλα αυτά είναι προς το συμφέρον των γειτονών μας αλλά βοηθούν και τη δική μας ενημεριακή ασφάλεια. Σήμερα θεωρώ ότι υπάρχει ένας κίνδυνος σε σχέση με τα ε, όσα να έχουμε μάθει από την Αραβική Άνοιξη. Μιλούμε για ενδιαφέροντα και αξίες ως αντιτιθέμενα πράγματα. Δεν θεωρείτε ότι οι αξίες της ε, πολιτικής γειτονίας ε, θεωρείτε ότι είναι κατά των συμφερόντων μας. Επίσης αναφέρατε το τρίγωνο το ρόλο των γειτόνων των γειτόνων και των εταίρων των εταίρων. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτούς τους παράγοντες, τους ιδιωτικούς παράγοντες που είναι πάρα πολύ βασικοί για την υλοποίηση των στόχων μας. Πώς νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να καλύψει τον ρόλο αυτών των παραγόντων στην ε, περιοχή μας. Ευχαριστούμε κύριε Κριστέα. Κίτσουκ. Κύριε Κρομάτσκι, έχουμε τρεις ομάδες χωρών. Η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία πρέπει να βελτιώσουν τη, τα δημοκρατικά δικαιώματα και να πλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει η ε, δημιουργία πλήρων περιοχών ελευθερών εμπορίου. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την συνεργασία μας με τις χώρες αυτές σε όλους τους τομείς. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε χώρες όπως η Αρμενία που είναι τμήμα της Ευρωασιατικής Οικονομικής Ένωσης και την Λευκορωσία. Εγώ δεν θα έβαζα το Αζερβαϊτζάν σε αυτές τις δύο χώρες. Για μένα είναι μια από τις πιο σημαντικές εταιρικές χώρες. Ο, το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι έχει πιο σημαντικό ρόλο με την ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άποψη αυτή θα ήθελα να ρωτήσω πώς θέλετε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με την Αρμενία και την Λευκορωσία και τι βήματα θα πρέπει να γίνουν για να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Τροχιά. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει μια ειδική αντιμετώπιση προς το Αζερβαϊτζάν για να συμμετοτέχει στην Ενεργειακή Ένωση και θέλετε να ακολουθήσει τα βήματα της Γεωργίας Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Και τέλος προς τον κύριο Μαζέν. Η περαιτέρω χρηματοδότηση για διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο στις νότιες όχθες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Μεσογείου μάλλον θα βοηθήσει την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της Ισλαμοφοβίας. Κύριος Παντζέρη, πολύ σύντομος πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να μας πούν κάτι προσκεκλημένοι μας, αφού τους ευχαριστήσω, να μας πούν πρώτα πρώτα το εξή. Θεωρείτε ότι υπάρχει σήμερα ισορροπία μεταξύ της ε, πολιτικής δυνήτησης προς Ανατολός και προς Νότον. Γιατί εγώ τώρα θεωρώ ότι υπάρχει ανισορροπία. Μεγάλο ενδιαφέρον προς Ανατολάς και πολύ λίγο προς Νότον. Προς Νότον νομίζω ότι στρέφεται κατά κάποιο τρόπο ε, σε σχέση με τον ε, κίνδυνο της τρομοκρατίας. Δεύτερη ερώτηση. Οι δυσκολίες της πολιτικής δυναμίας έχουν να κάνουν με την σημερινή ε, αδυναμία της εξωτερικής μας πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις γεωπολιτικές προοπτικές ολόκληρων περιφερειών και τις αντίστοιχες στρατηγικές και αυτό το διαπιστώσαμε με την πρόσφατη πολιτική γετνίαση, η οποία πηγαίνει από μια μεριά για ανάπτυξη και ανθρωπιστική ε, βοήθεια και από την άλλη μεριά ε, στην πολιτική αντίληψη κάποιων κράτων μελών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει κάποια πολιτική ισορροπία για να υπάρχει μια τέτοια πολιτική ε, που να συνάδει προς την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίασης, εντάξει δεν θέλω τώρα να, να σας πω το πώς θα αξιολογήσουν την αιρεσιμότητα. Είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε στο γόνατο ένα σχεδιασμό, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες μπορούν να διέπονται από αυτή την πολιτική. Να, α πούμε, μου δώσουν 10 ευρώ. 10 ευρώ να ξοδέψω αυτή την πολιτική, θα το κάνω, ούτω ώστε να βοηθήσω την πολιτική σταθερότητα τη νησία, γιατί είναι σημείο αναφορά για όλη την περιοχή. Απ' την άλλη μεριά, να δώσουμε από λίγο σε όλου, αυτό δεν πρόκειται να αντιστοιχεί σε κάποιο λογικό κριτήριο, ούτε θα λύσει κανένα πρόβλημα. Περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε, συναδελφέ Παντσέρη. Δεν ξέρω, ίσως δεν ξεγνωρίζετε ότι είναι ο κύριος Παντσέρη εκείνος που έχει αναλάβει την έκθεση για την κατάσταση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε όλες τις άλλες χώρες και κυρίως στις χώρες της, ε, ε της πολιτικής Επομένως είναι σημαντικά αυτό απαντήσετε και συμφωνεί ο κ. Παντσέρη. Οπότε πρώτα πρώτα λάβετε εσείς το λόγο, τρία λεπτά ο καθένας και κατόπιν ο εισηγητής μας ο Έντουαρτ και κατόπιν εγώ θα ολοκληρώσω. Πολύ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο ε, Τρομάτσκι. Είπατε, λέει ο κύριος Γκάλερ, ότι η Ρωσία ανέκαθεν ήταν αντίθετη με την προσέγγιση των χωρών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τον ΝΑΤΟ μόνο. Διάβασα ένα άρθρο της Frankfurt Allgemeine 10 Δεκεμβρίου του 2004 και λέει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν εκφράστηκε υπέρ, ε, ε, ε σχετικά μάλλον με μια ε, μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από συνομιλία με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σαπατέρο στη Μόσχα είπε ότι μέχρι και θα καλωσόριζε την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10-12 του 2004, πριν από 10 χρόνια και κάτι. Γιατί άλλαξε γνώμη η Μόσχα. Αυτό μήπως έχει λιγότερη σχέση με εμά και περισσότερο με τις εσωτερικές εξελίξεις της εσωτερικής πολιτικής στη Μόσχα, στη Ρωσία. Μήπως ε, ουσιαστικά αυτό κρύβεται πίσω από την πρίμνα που ανέκρουσε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρομάτσκι. Very briefly. Πάρα πολύ σύντομα. Κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα. Πώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας Ανέφερα ήδη το θέμα της σταθεροποίησης της Ουκρανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους επόμενους μήνες και χρόνια. Όχι μόνο η Ουκρανία. Και η Μολδαβία. Και η Γεωργία. Πρέπει να εστιάσουμε στις χώρες αυτές. Πρέπει να υπάρξει μια κάποια ισορροπία μεταξύ της ρωσικής ε, πολιτικής εναντίον των χωρών αυτών και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πώς μπορούμε να διαρθώσουμε σε ομάδες αυτές τις έξι χώρες. Βλέπω ότι υπάρχουν για μένα δύο ομάδες. Είπατε ότι η Μπελαρούς θα πρέπει να πάει μαζί με την Αρμενία γιατί είναι τμήμα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Μαζί με τη Ρωσία και το Καζακστάν. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κενό που κάμισο η Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσει αυτή η Ένωση. Δεν έχω βέβαια χρόνο να σε εξηγήσω γιατί. Το πρόβλημα του Αζερβαϊτζάν είναι απλό. Είναι μια χώρα που είναι μη δημοκρατική και αυταρχική. Ο πρόεδρος Αλίγεφ δεν ενδιαφέρεται σε να γίνει η δημοκρατικοποίηση του Αζερβαϊτζάν δεν ενδιαφέρεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα περιλαμβάνουν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων. Ενδιαφέρεται βέβαια για μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μόνο οικονομικό επίπεδο. Είναι καλό για αυτόν. Τον ενδιαφέρει αλλά δεν θέλει μια συνεργασία που θα βασίζεται στους δικούς μας κανόνες και στις δικές μας αξίες. Μια τελευταία παρατήρηση για τη θέση της Ρωσίας έναντι των χωρών της ε, Ανατολικής Γειτονίας. και την πολιτική στενότερων σχέσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πιστεύω ότι η πολιτική του Πούτιν ήταν ήδη μια πολιτική προσέγγισης κατά της προσέγγισης των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει άποψη τα τελευταία δέκα χρόνια. Όπως όμως είπα προηγουμένως στην παρουσίασή μου, πιστεύω ότι η ρωσική πολιτική ελίτ θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει μέλλον και έχουν αλλάξει το 2013 την άποψή τους και τώρα βλέπουμε ότι είναι και πάλι είναι πιο ανοιχτή σε καλύτερες σχέσεις των χωρών της ε, Ανατολικής Γειτονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριο Μάζεν τα τελευταία του σχόλια, παρακαλώ. Ταχυτερότερα. Ε, Δέθη ένα ερώτημα για τα συμφέροντα και τις αξίες. Είναι συμβατά αυτά, είναι αντικρουόμενα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε, οι ιδεαλιστές μπορεί να θεωρούν ότι καμιά φορά αυτά συγκρούονται, αλλά πάντα υπάρχει τρόπος να βρεθεί ένας ε, δρόμος, μια μέση εδώ. Είναι αξία η προώθηση της δημοκρατίας και υπάρχουν ε, πολλά να προτείνει κανείς και δεν είχα το χρόνο να το πω. Ένα σύντομο δίδαγμα ε, της Αραβικής Άνοιξης είναι ότι η δημοκρατία θέλει χρόνο και οι θεσμοί θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορούν να γίνουν ελεύθερες ε, εκλογές ε, χωρίς να υπάρχει μια σωστή φορευτική επιτροπή. Και όλες οι χώρες είχαν πρόβλημα με αυτό. Και το κοινοβούλιο είναι πάντα ένα αποτελεσματικό εργαλείο ε, δημοκρατίας, αλλά όταν ε, υποχρηματοδοτείται ένα κοινοβούλιο και υποστελεχώνεται, υπολειτουργεί κιόλας. Υπάρχουν προτεραιότητες, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο και πώς βοηθάει στην καταπολέμηση τρομοκρατίας και βεβαίω βοηθά. Στην περιοχή πολύ ριζοσπαστικοποιήθηκαν λόγω των στρεβλών ιδεών για το τι εστί Δύση, η Δυτική Ευρώπη και πώς μεταχειρίζεται τους μουσουλμάνους. Δεν έρχονται στην Ευρώπη, δεν ξέρουν, δεν βλέπουν ευρωπαϊκή τηλεόραση, ακούνε μα, δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ. Ε, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου και τους ριζοσπαστικοποιούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Για το θέμα της ασφάλειας επιτάχυνση της υποστήριξης της ε, ε, αντιμετώπισης του θέματος των προσφύγων. Είναι κρίσιμο αυτό. Παντού στην περιοχή. Και όχι μόνο στην Ιορδανία ή το Λίβανο κατά τα άλλα. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, είναι πρόσφυγες. Τους έχω δει και στο Κάιρο. Είναι άστεγοι, ε, ζήτια ανέβουν, δεν έχουν τι να κάνουν. Ε, και αυτό είναι μια επένδυση στην ασφάλεια αν αντιμετωπιστεί το θέμα των προσφύγων. Και για τους ελέγχους στα σύνορα χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και πιο αποτελεσματική και των αντιστοίχων ε, αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμων μας και τον κύριο Γκρομάτσκι και τον δόκτωρα Μάζεν. Ε, πολύ χρήσιμη ανάλυση τους ε, το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει και να μεταρρυθμίσει πολιτική γειτονία της. Ε, ακούσαμε και τη δική σας ανάλυση και τη μελέτη σας και με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσουμε και την ανάλυση για την νότια γειτονία. Ζητώ συγγνώμη στον εισηγητή μας Έντουαρτ Κούκαν για τους χρονικούς περιορισμούς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω παρόλα αυτά να είχαμε πολύ γόνιμη συζήτηση και επικοδομητική. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι η πρώτη συζήτηση της έξω του κ. Κούκαν έχει προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Απριλίου Αργότερα θα συζητήσουμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες. Για τα διάφορα δεν πιστεύω να θέλει κανείς άλλος να προσθέσει και με την άδεια του Προέδρου να πω ότι στις 9 Μαρτίου είναι επόμενη συνεδρίαση, 7 η ώρα στο Στρασβούργο. Διακόπτεται η συνεδρίαση, λίγοι δηλαδή, και ε, όσοι θέλουν να παραμείνουν για το διευρυγμένο Προεδρείο, όσοι πρέπει δηλαδή να παραμείνουν, οι υπόλοιποι, καλό σας βράδυ, σχολάσατε.